Ίσως να είναι αποτέλεσμα της κρίσης, ίσως όχι, αλλά γεγονός είναι πως σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει πολλές τέτοιες απαιτήσει. Και βεβαίω οποιαδήποτε νέα αγορά ανέρχεται αντιγράφει και αυτή την ίδια στρατηγική. Γιατί, ναι, αυτό μπορεί να εφαρμοστεί ίσως σε μια χώρα όπως η Βραζιλία ή η Κίνα ή ίσως και η Ινδία, αλλά δεν μπορεί να λειτουργήσει στην Νότια Αφρική μια χώρα μεσαίου μεγέθους ή μια χώρα μικρού μεγέθους. Οπότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Επίσης, αν δείτε τα φωτοβολταϊκά, και εκεί πέρα υπάρχει απέτηση για τοπικό ποσοστό παραγωγής και άλλη μια εξέλιξη που έχει καταγραφεί στην αγορά είναι η αύξηση των ε, εμπορικών ε, διαμαχών, το αντι-dumping κτλ. Οι τρεις τελευταίες διαφάνειες λοιπόν είναι αποδείξεις από την αγορά πως τα πράγματα πηγαίνουν προς τη λάθος κατεύθυνση και υπάρχει μια τάση λανθασμένη. Εάν δηλαδή είναι κανείς μια εταιρεία φαντάζεστε πώς μπορεί να κάνει επενδύσεις με αυτό το μοσαϊκό κανόνων που υπάρχει. Γιατί είναι προβληματικό αυτό. Είναι προβληματικό γιατί η βιομηχανία αυτή τη στιγμή ανταγωνίζεται με άλλες ενεργειακές τεχνολογίες και στην αγορά. Το μόνο θέμα είναι το κόστος της ενέργειας. Αν δείτε το γράφημα αυτό βλέπετε πως τα φωτοβολταϊκά και κάπως τα αεολικά έχουν μειώσει το κόστος τους σημαντικά τα τελευταία χρόνια εάν είχαμε ένα πιο μακροπρόθεσμο σχεδιάγραμμα θα βλέπαμε κάπου και την αιωλική ενέργεια. Αλλά υπάρχει βεβαίως πολύ, υπάρχουν πολλά μέταλλα στον εξοπλισμό αυτό, το κοστίζει, αλλά μπορεί να μειωθεί. Βλέπετε πως ε, η αιωλική αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν ανταγωνιστική με κάποια ορυκτά καύσιμα σε πολλά μέρη του κόσμου. Και επίσης ε, μειώνεται και γρήγορα η τιμή. Αυτό είναι μια συμφωνία που θα ήθελε η βιομηχανία να κάνει με τους πολιτικούς, ότι δηλαδή ναι μπορούν να δώσουν χαμηλό κόστος αγοράς αρκεί να συνεχίσουν να αυξάνονται οι αγορές αυτές. Οπότε αν πάμε προς την άλλη κατεύθυνση προς μια πανεθνικοποίηση, τότε μπορώ να σας πω πως θα αναστραφεί αυτή η τάση και αυτό θα είναι προβληματικό για τον κλάδο. Γι' αυτό θεωρεί ο κλάδος πως η πρωτοβουλία ΑΠΕΚ είναι πάρα πολύ καλή. Είναι κάτι το θετικό. Και θα επανέλθουμε στο πόσο θετικό είναι, αλλά σε ένα γενικό επίπεδο είναι καλό να βλέπουμε όπως ε, και αυτή η περιοχή του πλανήτη ε, εμπλέκεται γιατί είχαν ε, εμπλακεί στις συνομιλίες του ΠΟΕ για τις περιβαλλοντικές υπηρεσίες. Θα το πει και ο Άλφος. Επίσης βλέπουμε κάποιες εξελίξεις στις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου που επίσης έχουν απασχολήσει το τη βιομηχανία. Δηλαδή θα σχηματιστεί μια κρίσιμη μάζα και θα είναι μετά πάρα πολύ εύκολο να περάσουμε στο επόμενο επίπεδο. Είτε σε μια τριμερή είτε σε μια πολυμερή συμφωνία. Οπότε έχουμε πιθανώς μια καλή εξέλιξη. Αλλά το θέμα είναι πώς θα το επιταχύνουμε. Δεν μπορούμε να περιμένουμε 12 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να εκμεταλλευτούμε τις εξελίξεις αυτές και γιατί η βιομηχανία ε, αντιμετωπίζει κρίση. Αν δούμε λοιπόν τη λίστα του ΑΠΕΚ και πλησιάζω τώρα προς το τέλος. Πολιτικά μιλώντας είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Αν δούμε τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Είναι 54, 54 υποκεφάλαια με ένα 5% maximum. Κάτι το οποίο βέβαια θα μπορούσε να είναι ένα 70% του παγκοσμίου εμπορίου. Κάτι το πάρα πολύ θετικό από την πλευρά του ΑΠΕΚ. Και αν μπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα καλύψουμε το 95%. Αλλά το πρόβλημα με το ΠΕΚ είναι πως είναι πως δεν είναι μεγάλη η δέσμευση. Πολλές από τις χώρες περιοχής έχουν ε, δασμούς κάτω από το 5%. Δεν είναι λοιπόν φοβερά μεγάλη αυτή η δέσμευση και αν ε, ρωτήσουμε τη βιομηχανία θα ήθελαν ίσως μια άλλη πρωτοβουλία. Και αυτό πρέπει να δει η Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα ενθαρρύνει τις θετικές εξελίξεις που έχουν ξεκινήσει στην ΑΠΕΚ και να πάμε παραπέρα. Επίσης η πρωτοβουλία αυτή δεν αντιμετωπίζει τις μη δασμολογικούς φραγμούς, αυτά περί τοπικής παραγωγής κτλ. Οπότε πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να διευρύνει και να εμβαθύνει σε σχέση με το που είμαστε τώρα και αναμένω κάποιες από τις συζητήσεις που θα έχουμε στο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει αυτό. Και οπωσδήποτε παραλαμβάνω το επιχείρημά μου. Βλέπω και την ε, διατλαντική συνεργασία ως ένα δυνητικά σημαντικό μέσο έτσι ώστε όλα, όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να γίνει μια σχεδόν ε, παγκόσμια συμφωνία. Και πριν κλείσω, να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν μιλάμε για τοπικό περιεχόμενο, κάποιοι θεωρούν πως είναι μια έξυπνη βιομηχανική πολιτική για να υπάρξει κάποια τοπική παραγωγή, τοπικές δουλειές, αλλά γεγονός είναι πως η τοπική παραγωγή ε, είναι στο DNA αυτών των τεχνολογιών. Εδώ έχουμε ένα παράδειγμα από τον αιωλικό τομέα, όπου βλέπουμε την αλυσίδα αυτή, όπου ε, εξορισμού η συντήρηση και η απόσυρση και όλα αυτά είναι εξορισμού τοπικά. Αλλά βέβαια η κατασκευή κτλ. είναι εισαγόμενα. Αλλά και αυτό εξαρτάται από το μέγεθος της αγοράς. Έτσι. Δυνητικά Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνονται σε τοπικό επίπεδο. Το θέμα είναι πως ούτως ή άλλως θα υπάρξει αρκετά μεγάλη τοπική συμμετοχή και στον τομέα των φωτοβολταϊκών. Δίνεται έμφαση στα πάνελ που εισάγουμε από την Κίνα. Δεν συζητάμε τις δουλειές που υπάρχουν ε, στον τομέα της εγκατάστασης και της συντήρησης. Δεν μιλάμε για τις ε, εταιρείες ε, υψηλής προσθέμενης αξίας ε, που κάνουν την έρευνα. Οπότε δεν είναι ότι όποιος κερδίζει κάτι το αφαιρεί από κάποιον άλλον, όχι μπορούμε όλοι να κερδίσουμε. Θα σταματήσω εδώ. Σας παρακαλώ λοιπόν βοηθήστε μας να έχουμε ίσους όρους ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο το στομότερο δυνατόν να εκμεταλλευτούμε τα επόμενα χρονιά για να το εξασφαλίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενη ομιλήτρια, η κυρία Μότα, αλλά αναπληρώτρια Γενική Διευθυντή στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Που βρίσκεστε, ο... έχετε το λόγο για 12 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ για να σας μιλήσω για τις διαπραγματεύσεις που λαμβάνουν χώρα στον ε, Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου και τις εξελίξεις που έχουν λάβει η χώρα πρόσφατα και πώς αυτές σχετίζονται με το τι προσπαθούν να επιτύχουν οι χώρες σε παγκοσμίο επίπεδο. Να σας περιγράψω λιγάκι το πλαίσιο αυτής της διαπραγμάτευσης στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Οι συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα εκεί για τα περιβαλλοντικά αγαθά και τις υπηρεσίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Πρόκειται για την πρώτη φορά που περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις έχουν ξεκινήσει υπό την αιγίδα του πολυμερού συστήματος εμπορίας και πρέπει να αντιληφθούμε τη σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος βάσει των κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου όταν δημιουργήθηκε το ΓΚΑΤ το 1947 και όταν ακολούθησαν άλλες συμφωνίες όπως η Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες για τους φραγμούς στο εμπόριο οι χώρες δημιούργησαν για τους αυτούς τους χώρο περιβαλλοντικό δηλαδή δημιούργησαν περιθώριο αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζητημάτων στο πλαίσιο διεθνών κανόνων εμπορίου. Ωστόσο αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Πολυμερού συστήματος εμπορίας όπου έχει ξεκινήσει διαπραγμάτευση με συγκεκριμένο περιβαλλοντικό στόχο. Αυτές λοιπόν οι διαπραγματεύσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές. Δεν ξεκίνησαν επιμέρους, απομονωμένες, ε, εντάσσονται στο πλαίσιο ενός πακέτου ζητημάτων. Το περιβαλλοντικό λοιπόν κεφάλαιο του γύρου τη στόχας συνίσταται στην εξέταση τη σχέση μεταξύ κανόνων του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου και των Διεθνών Περιβαλλοντικών Συνθήκων συνίσταται στην εξέταση του ζητήματος των ε, αλληλευτικών επιχορηγήσεων και του κατά πόσο κάποιες χώρες ε, επιδοτούν υπερβολικά τους αλληλευτικούς τους τομείς με αποτέλεσμα την ε, εξάλληψη των ηχθιαποθεμάτων. Και το άλλο κομμάτι είναι αυτό που θα δούμε σήμερα, την απελευθέρωση του εμπορίου για περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίες. Κατά την άποψή μου πρέπει οπωσδήποτε να επιτύχει αυτή η πρώτη στην ιστορία διαπραγμάτευση, περιβαλλοντική διαπραγμάτευση υπό την αιγύδα του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Η λογική στην οποία βασίζεται αυτή η διαπραγμάτευση είναι σαφής. Δεν έχει νόημα ο κόσμος να τιμωρεί τεχνολογίες που προστατεύουν το περιβάλλον. Ειδικότερα λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική κρίση που έχουμε σήμερα. Δεν χρειάζεται να αυτομαστιγωνόμαστε προς μην επιτρέποντα τι τεχνολογίε αυτέ να διέρχονται τα σύνορα και να έχουν πρόσβαση σε αυτέ όσοι τι χρειάζονται. Η λογική λοιπόν είναι πολύ απλή. Πρέπει να μπορούν να ταξιδέψουν αυτά τα αγαθά και αυτέ οι υπηρεσίε. Το περιβάλλον δεν γνωρίζει σύνορα. Κατά την άποψή μου, Δυστυχώ, όταν ξεκίνησε το περιβαλλοντικό κεφάλαιο του γύρου τη Δόχα, μαζί με τη διαπραγμάτευση για τα αγαθά και τι υπηρεσίε, η κοινωνία των πολιτών που είχε πίεση τόσο πολύ για αυτέ τι διαπραγματεύσει, διαπραγματεύσεις σχεδόν τις εγκατέλειψε. Για χρόνια ακούγαμε ατελείωτες συζητήσει για το πόσο ήταν απολύτως απαραίτητο το greening, ότι ο Διεθνής Οργανισμός Εμπορίου έπρεπε να ευαισθητοποιηθεί από περιβαλλοντική άποψη και αυτή τη στιγμή ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις αυτές. Μας εξέπληξε το γεγονός ότι η κοινωνία των πολιτών αποσύρθηκε και άφησε τις διαπραγματεύσεις στο ελαιός των χωρών. Μόνο σε έναν τομέα δραστηριοποιήθηκε η κοινωνία των πολιτών στις αλληλευτικές επιδοτήσεις, όπου πολλοί εξειδικευμένες μη καπαό παρενέβησαν, αλλά σε όλους τους άλλους τομείς των διαπραγματεύσεων η κοινωνία των πολιτών εγκατέλειψε τις διαπραγματεύσεις. Κατά την άποψή μου είναι εύκολο να ορίσουμε την επιτυχία αυτής της διαπραγμάτευσης. Εσεί, τα μέλη του Κοινοβουλίου, θα έχετε ακούσει ένα σώρο διαφορετικέ προσεγγίσεις στη Γενέβη. Μια προσέγγιση βάση έργων, μια προσέγγιση βάση λίστα. Διάφορε τέτοιε προσεγγίσει, αλλά εν τέλει, ανεξαρτήτω τη αρχιτεκτονική που θα υιοθετηθεί και τη οδού που θα επιλεγεί για αυτέ τι διαπραγματεύσει κατά την απόψή μου, η επιτυχία μπορεί να μετρηθεί με σαφή τρόπο. Το πρώτο μέτρο επιτυχίας βασίζεται στον αριθμό στο πλήθο προϊόντων για τα οποία θα απελευθερωθεί το εμπόριο. Εν τέλει μιλάμε για προϊόντα που διέρχονται συνόρων και το πόσο εύκολο είναι για αυτά. Όσο μεγαλύτερη είναι η λίστα των εν λόγω προϊόντων, τόσο πιο επιτυχής θα είναι η διαπραγματεύση. Τώρα φυσικά πρέπει να υπάρχουν ισχυρέ, προποθέσει και κριτήρια για περιβαλλοντική φύση για αυτά τα προϊόντα. Το δεύτερο κριτήριο επιτυχίας είναι το πλήθο των χωρών που θα συμμετέχουν στη συμφωνία. Όσο περισσότεροι παίκτες υπάρχουν για την απελευθέρωση των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών, τόσο καλύτερο θα είναι το περιβάλλον. Και το τρίτο και τελευταίο κριτήριο, κατά την άποψή μου, είναι η δεσμευτική φύση της συμφωνίας που θα επιτευχθεί. Εάν ε, επιτύχουμε ένα χαλαρό πλαίσιο, το αποτέλεσμα θα είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με εκείνο μια δεσμευτική συμφωνία, ενό δεσμευτικού μηχανισμού. Και κάποιοι από εσά θα έλεγαν τι κάνουμε με τι ανάγκε των αναπτυσσόμενων χωρών όσον αφορά τη μέτρηση τη επιτυχία αυτή των διαπραγματεύσεων. Πιστεύω ότι οι ανάγκε των αναπτυσσόμενων χωρών μέσω αυτών των διαπραγματεύσεων θα εξαρτηθούν και αποτελούν συνάρτηση του βαθμού δεσμευσή του. Εάν οι αναπτυσσόμενε χώρε δεν προωθήσουν λίστε προϊόντων που τι ενδιαφέρουν οικονομικά και περιβαλλοντικά, τότε αυτέ οι διαπραγματεύσει δεν θα του είναι ιδιαίτερα ωφέλιμε. Ο βαθμό, λοιπόν εμπλοκή του θα αποτελέσει παράγοντα κλειδί, καθοριστικό παράγοντα για το πόσο θα υποφεληθούν αυτών των διαπραγματεύσεων. Τι θα κερδίσουν από αυτέ τι διαπραγματεύσει. Τώρα το ερώτημα που προφανώ έχουν όλοι στο μυαλό του, είναι πώ είπε και κατάφερε να επιτύχει όσα έκανε ενώ καθυστερούν ταυτόχρονα οι διαπραγματεύσει του Παγκόσμιου ε, Οργανισμού Εμπορίου για τόσο καιρό στη συμφωνία ΑΠΕΚ συμβαίνει κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί για πολλά χρόνια. Συνεργασία μεταξύ ΕΠΑ και Κίνας. Καθίσαν γύρω από το τραπέζι διαπραγματεύσεων και κατάφεραν να συνάψουν, να καταλήξουν σε μια συμφωνία μετά από πολλά χρόνια. Στην ΕΠΑΚ. Πέτυχαν θα έλεγε κανείς γιατί είναι λιγότεροι οι συμμετέχοντες. Άλλοι μπορούν να πούν ότι μιλάμε για λιγότερα προϊόντα από ό,τι αυτά που εξετάζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου. Άλλοι θα έλεγαν ότι η ΕΠΑΚ είναι λιγότερο πολιτικοποιημένο φόρουμ σε σχέση με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Ίσως όλα αυτά έκαναν τις διαπραγματεύσει στην ΑΠΕΚ πιο εύκολη. Εγώ πιστεύω κάτι διαφορετικό από όλες αυτές τις θεωρίες. Πιστεύω ότι στην ΕΠΑΚ κατάφεραν να επιτύχουν συμφωνία, γιατί αυτή η συμφωνία είναι μη δεσμευτική. Μόλις πάψει να είναι δεσμευτική μια συμφωνία, είναι πολύ εύκολο να συμφωνήσει κανεί να συμμετέχει. Είναι πολύ πιο, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσει κανεί να συμμετέχει δεσμευτικά αύριο. Και το ερώτημα είναι πώ θα επιτύχουν μια τέτοια δεσμευτική συμφωνία. Το ζήτημα τώρα είναι ότι ο κόσμο πρέπει να αποφασίσει τι περιβαλλοντικέ τακτικέ θέλει να ακολουθεί και τι ε, περιβαλλοντικό εμπορικό κανόνα. Ε, νομοθεσία θέλει να ακολουθεί. Θέλουμε ισχυρή νομοθεσία ή όχι. Κατά την άποψή μου πρέπει οπωσδήποτε να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις πολυμερός στον Παγκοσμίο Οργανισμό Εμπορίου. Όχι μόνο γιατί είναι η πρώτη διαπραγμάτευση περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αλλά και γιατί χρειάζεται να συνεχίσουμε να οικοδομούμε δεσμευτικά εμπορικούς κανόνες, βάσει εμπορικών κανόνων που έχει καθιερώσει ο Παγκοσμίος Οργανισμός Εμπορίου. Πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το κεκτημένο και να το εξελίξουμε Πρέπει να βασιστούμε σε εμπορικούς κανόνες που υπάρχουν, που εργάστηκαν κάποιοι σκληρά για να τους δημιουργήσουν. Η Συμφωνία ΕΠΑ, κατά την άποψή μου, αποτελεί σημαντικό ορόσημο, καθώς κινούμαστε προς μια πολυμερή συμφωνία. Και κατά την άποψή μου, σε διεθνές επίπεδο, πρέπει να αρχίσουμε να οικοδομούμε πάνω σε αυτή τη Συμφωνία ΕΠΑΚ. Αυτή η λίστα περιλαμβάνεται από 54 προϊόντα. Αυτά είναι μερικά μόνο από τα 400 ουσιαστικά που υπάρχουν στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί εύκολα να συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία ΕΠΑΚ, διότι ουσιαστικά όλα οι δασμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτω του 5% για όλα αυτά τα προϊόντα που βρίσκονται στη λίστα. Δεν χρειάζεται λοιπόν καμία προσαρμογή για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, η συμμετοχή τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη συμφωνία είναι σε τεράστιο βαθμό συμβολική. Διευρύνει τη συμφωνία, δίνει ορμή σε μια πολύ μεγαλύτερη συμφωνία και επίση θα προσελκύσει σιγά σιγά τι περιβαλλοντικέ υπηρεσίε που άφησε πίσω η ΕΠΑΚ. Διότι πρέπει να θυμόμαστε ότι οι διαπραγματεύσει του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου δεν αφορούν μόνο τα αγαθά, αλλά και τι περιβαλλοντικέ υπηρεσίε. Θα μπορούσε επίση να προσελκύσει ε, να, να φέρει μεγαλύτερη επιτυχία στις γενικότερες περιβαλλοντικές διαπραγματεύσεις. Για μένα το κύριο μάθημα είναι ότι υπάρχουν αντισταθμιστικές συνθήκες. Μπορούμε να έχουμε μία λιγότερο φιλόδοξη συμφωνία που θα είναι δεσμευτική, μια περισσότερο φιλόδοξη που δεν θα είναι δεσμευτική. Τι από τα δύο θα πρέπει να επιλέξουμε. Θα πρέπει να κάνουμε υποχωρήσεις όσον αφορά το δεσμευτικό το εύρο τη συμφωνία ώστε να επιτύχουμε δεσμευτική συμφωνία. Αυτό θα ήθελα να σκεφτείτε όλοι. Θα ολοκληρώσω με δύο περαιτέρω μηνύματα. Το πρώτο είναι ότι σήμερα γίνονται αυτές οι διαπραγματεύσεις σε τελείως διαφορετικό επίπεδο από τότε που ξεκίνησαν. Σήμερα υπάρχει τεράστια τριβή μεταξύ του τομέα του εμπορίου και του τομέα του περιβάλλοντος, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι οι κλιματικές διαπραγματεύσεις διεθνώς έχουν παραμείνει στάσιμε και αυτό το αδιέξοδο αυτών των διαπραγματεύσεων επηρέασε τις διαπραγματεύσεις των Διεθνή Οργανισμών Εμπορίου. Διαρκώς αυξάνονται οι εντάσεις μεταξύ χωρών για θέματα όπως ο φόρος άνθρακα, η επισήμανση του άνθρακα, πώς, το πώς κατανέμονται οι αντισταθμίσεις στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας και διενέξεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου, όπου κάποιες χώρες αμφισβητούν τις επιδοτήσεις που κάποιες άλλες δίνουν στους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και το θέμα των τοπικών απαιτήσεων περιεχομένου. Το να πετύχουμε μια συμφωνία περιβαλλοντικού αγαθών είναι συμβολικό σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να αγκαταλείψουμε τις τριβές και να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε. Μια τέτοια συμφωνία για τα περιβαλλοντικά αγαθά βάσει αυτή τη λίστα που εξετάζεται αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου ε, θα περιλαμβάνει πολλά προϊόντα που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των κλιματολογικών αλλαγών. Το τελικό μήνυμα που θέλω να πω είναι ότι σήμερα έχουμε καθολικές αλυσίδε αξιών όσον αφορά το εμπόριο. Δηλαδή τα προϊόντα δεν παράγονται μόνο σε μία χώρα Α και δεν εξάγονται μόνο σε μία χώρα Β. Παράγονται σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ένα ηλιακό συλλέκτη, ακόμη και αν γράφει πάνω Made in China, ουσιαστικά πολλά ε, εξαρτήματά του έχουν ε, κατασκευαστεί στη Γερμανία, στις ΗΠΑ και έχουν σταλεί στην Κίνα για συναρμολόγηση και μετά επανασταλεί για πώληση. Συνεπώ, οι δασμοί σήμερα έχουν πολύ λιγότερο νόημα από ό,τι παλιότερα. Δεν είχαν νόημα ούτε παλιότερα, αλλά σήμερα δεν έχουν θέση σε έναν ε, κόσμο ο οποίο ενοποιείται όλο και περισσότερο. Και αυτό ισχύει ειδικότερα στον περιβαλλοντικό τομέα, ο είναι εξαιρετικά δυναμικό και θα ήταν κρίμα να συνεχίσουμε να έχουμε αυτού του δασμού τόσο από εμπορική όσο και από περιβαλλοντική άποψη. Κατά την άποψή μου. Ευχαριστώ. Thank you very Next. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή ο κύριος Βαν Σλάτεν Διευθυντής της Βιομηχανικής Πολιτικής ε, της Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χημικής Βιομηχανίας, του ΣΕΦΙΚ. Έχετε το λόγο. 12 λεπτά κατά τώρα και σας ευχαριστούμε που εδώ. Κύριε Πρόεδρε, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο που κάλεσε την ΣΕΦΙΚ σε αυτή την ακρόαση. Η πρόταση να διαγραφούν για η τελωνιακή δασμή, για τα πράσινα ή περιβαλλοντικά αγαθά είναι της μόδας και όλοι θέλουν πραγματικά να καταλήξουμε σε μια κατάσταση στην οποία οι πάντες θα κερδίσουν και θα, προς το καλό της οικονομίας, του περιβάλλοντος και για κοινωνικούς λόγους. Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είπε ότι περαιτέρω πρόοδος απαιτείται προς την απελευθέρωση της, του εμπορίου των ε, περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Η χημική βιομηχανία πιστεύει στο ελεύθερο εμπόριο και είναι υπέρ της ε, περαιτέρω ε, απελευθέρωσης στα πλαίσια πολυμερών ε, συμφωνιών, πολυπλών Ιδιαίτερος είναι υπέρ της ε, διαγραφής των διαφόρων τελωνιακών ε, τελών. Παρόλα αυτά, εξαιτίας κάποιων λανθασμένων αντιλήψεων και ορισμών, πιστεύουμε ότι κάτι τέτοιο δεν ε, έχει σταθερή βάση και έχει διάφορα προβλήματα. Η συζήτηση στον ΠΟΕ για την απελευθέρωση συνεχίζεται περίπου εδώ και 10 χρόνια, χωρίς να καταλήγει πουθενά. Ένας από τους λόγους είναι ότι τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να συμφωνήσουν στο τι είναι αυτά τα περιβαλλοντικά αγαθά. Και νομίζω ότι για να σας δείξω πόσο πολύπλοκο είναι θα σας μιλήσω με κάποια παραδείγματα. Το χλώριο χρειάζεται για την εξηγήση του πόσιμου ύδατος και έτσι με τον τρόπο αυτό σώζονται ζωή σε εκατομμυρίων ανθρώπων. Βεβαίω, αν δεν χρησιμοποιηθεί σωστά το χλώριο, μπορεί να είναι επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία. Καλή λόγη είναι το χλώριο ή όχι. Επίσης, ε, το βιοεθανόλη που γίνεται από ζαχαρότευτα Βραζιλίας είναι καλή, ενώ αυτή που γίνεται από τα ευρωπαϊκή παραλλαγή των ζαχαροτεύτλων είναι κακή. Τι θα πρέπει να κάνουμε τώρα, να θεωρηθεί η βιοεθανόλη ως περιβαλλοντικό αγαθό δεδομένου ότι έχει επιπτώσεις για τους για στα είδη διατροφής. Θα πρέπει η βιοεθανόλη να θεωρηθεί ε, λοιπόν ως θετική ή αρνητική. Επίσης, οι λαμπτήρες που περιέχουν ε, υδράργυρο είναι επιβλαβείς ή όχι. Καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές λαμβάνονται ε, αυθαίρετες αποφάσεις δεδομένου και κάποια θέματα, δεδομένου ότι το θέμα είναι πολύ πολύπλοκο. Το πρόβλημα του ορισμού επίσης ε, μας οδηγεί σε ένα άλλο θέμα που αφορά το εμπόριο, κυρίως αυτό των διακρίσεων που μπορούν ε, να ε, υποστούν κάποιοι εξαιτία των ορισμών, κυρίως όταν πρόκειται για θέματα που αφορούν το πρασίνισμα, το περιβάλλον, το φιλικό προς το κλίμα και τα προϊόντα τα, των ανάσημων πηγών ενέργειας. Οι προτάσεις επιτάπητος ε, ε, στη Γενέβη είναι μια αυθαίρετη συλλογή αγαθών που ε, υποκειμενικά θεωρούνται φιλικά προς το περιβάλλον, φιλικές προς το περιβάλλον. Και βεβαίως δημιουργούν διακρίσεις για κάποια άλλους λόγους, για άλλα προϊόντα. Ακόμη και το απορριπαντικό πολλές φορές που χρησιμοποιούμε είναι κάτι το οποίο ε, όταν χρησιμοποιείται σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ανάλογα με την αλλαγή του ε, θερμοκρασίες. Κατά συνέπεια θα πρέπει να διερωτηθούμε πραγματικά εάν οι διάφορες χώρες δεν θα πρέπει να κάνοντας αυτές τις μελέτες να δουν κατά πόσο το αρχικό προϊόν και όχι το τελικό είναι αυτό το οποίο επηρεάζει ε, τα πράγματα, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε αναπτυσσόμενε υποανάπτυξη χώρε. Όλες αυτές οι συζητήσεις μας οδηγούν επίση στο θέμα των ε, αλυσίδων αξιών και θα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικές είναι για την εμπορική πολιτική μιας χώρας. Άλλοι θα πούνε ότι θα πρέπει να απελευθερώσετε τα αρχικά προϊόντα δεδομένου ότι όσο περισσότερο ε, επεξεργάζεται κάποιος τα προϊόντα, καταλήξει σε τελικά προϊόντα, τόσο περισσότερο αυξάνεται η τιμή. Η Γερμανία, Φερρυπίν, είναι χώρα που παράγει πολυσιλικόνες, που είναι ένα βασικό υλικό για τα ε, ηλιακά κάτωπρα, για τους ηλιακούς συλλέκτες. Ενώ η Κίνα παράγει τους ηλιακούς συλλέκτες, εισάγοντας τα πολυσιλικόνες. Τελικά η έλλειψη σαφών ορισμών οδηγεί σε ε, προτάσεις οι οποίες είναι παράξενες. Όσον αφορά την ε, έννοια της ε, χρησιμότητας ή όχι κατάργησης των τελών για τα περιβαλλοντικά αγαθά. Τα αγαθά που χρησιμοποιούνται για περιβαλλοντικούς λόγους ε, πρέπει να πούμε ότι είναι περιβαλλοντικά, άρα να μην ε, τους επιβάλλονται τέλη. Πολλές φορές ξέρουμε ότι τέτοιου είδους προτάσεις τις ε, απορρίπτει η χημική βιομηχανία, δεδομένου ότι είναι από την άποψη της γραφειοκρατίας πάρα πολύ επαχθής και μπορούν να οδηγήσουν και σε φαινόμενα διαφοράς. Και επίσης θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το τελικό προϊόν. Δεν έχουμε κακά και καλά προϊόντα, αλλά πώς τα χρησιμοποιούμε. Και θα πρέπει να δούμε και για ποιους λόγους χρησιμοποιούνται. Το να, μπορέσουμε, το να εισαγάγουμε διαχωρισμούς μεταξύ καλών ή κακών προϊόντων, για τιμενικούς λόγους, μας ανοίγει δρόμους οι οποίοι δύσκολα μπορούν να ε, ακολουθηθούν και θα πρέπει να δούμε και για ή ηθικού λόγου πώς χρησιμοποιούν διάφορα προϊόντα. Παρ' όλα αυτά, εάν τα τέλη χρησιμοποιούνται για την ε, προώθηση κάποιων παρατηρήσεων ή ε, ηθικού περιεχομένου, θα πρέπει ε, τα τέλη λογικά να αυξηθούν τουλάχιστον σε ένα επίπεδο για, ο, που θα πρέπει να το ίδιο για όλα τα προϊόντα. Όσον αφορά την πρωτοβουλία της ΑΠΕΚ, είμαστε κατά και είμαστε κατά οποιασδήποτε πρωτοβουλίας της ΑΠΕΚ που θεωρείται ως περιβαλλοντική. Δεδομένου ότι θα πρέπει να δούμε τι ε, σημαίνουν όλα αυτά τα ενεργειακά περιβαλλοντικά αγαθά, ο κατάλογος αυτός των 54 προϊόντων και θα πρέπει να δούμε και τι σημαίνει η έννοια της ε, ενεργειακά αποδοτικής που χρησιμοποιείται. Μπορεί να μας οδηγήσει πολλές φορές σε προβλήματα. Δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με αυτή την ε, προοπτική και το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να προτείνουμε είναι η πρωτοβουλία αυτή για την προώθηση σε επίπεδο ΠΟΕ να γίνει ε, συμφωνία πολυμερής. Συμπερασματικά, για όλους αυτούς τους λόγους, η χημική βιομηχανία πιστεύει ότι θα ήταν καλύτερα εάν οι κυβερνήσεις έκαναν πολυμερείς ε, σοβαρές διαπραγματεύσεις για να μειώσουν ή να καταργήσουν όλες τις, ε, τα βιομηχανικά τέλη από όλα, για όλα τα προϊόντα αντί να αρχίσουν να ασχολούνται με ένα ε, θέμα που θα τους οδηγήσει σε αποτελέσματα αυθαίρετα και ποτέ δεν υπάρχει συμφωνία από ό,τι βλέπουμε. Μετά από 10 χρόνια στασιμότητα συζητή στη Γενέβη ε, καταλαβαίνετε ότι μπορούμε να πούμε ότι το όλο αυτό εγχείρημα είναι εθνησυγενές. Σύμφωνα με την μελέτη επιπτώσεων που έγινε το 2011 για την Επιτροπή, ε, τα ωφέλη από την απελευθέρωση των ε, περιβαλλοντικών αγαθών ε, μπορούν να αποφέρουν μόνο 2 εκατομμύρια δις, ενώ εάν αν έχουμε μια γενική συμφωνία. Αν έχουμε όμως τομεακές συμφωνίες χωριστέ, στον τομέα της χημίας, των εξοπλισμών και των ηλεκτρονικών θα μπορούσαμε να αυξήσουμε το ΑΕΠ κατά 17 δις δολάρια. Η χημική βιομηχανία λοιπόν είναι ε, υπέρ το να γίνει η, η απελευθέρωση τμηματικά. Στον τομέα των ε, χημικών προϊόντων η βιομηχανία έχει παρουσιάσει μια πρόταση ε, απελευθέρωσης των τελών σε επίπεδο ΠΟΕ, ε, την οποία πιστεύουμε ότι όλες οι μεγάλες χώρες, την οποία πιστεύουμε ότι όλες οι χώρες θα πρέπει να προσχωρήσουν. Πιστεύουμε ότι μόνον έτσι θα μπορέσουν τέτοιου είδους οικονομίες και επενδύσεις να έχουν θετικά αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Να ευχαριστώ. Θέλαμε και αυτή την άποψη βεβαίω. Τελευταίος ομιλητής Φάμπια Ντελκρός. Ε, αρμόδιος για σχέσεις με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για την General Electric. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε καθηγητά, εξ ονόματος των φίλων μου που βρίσκονται εδώ πέρα, ενώ βεβαίως την Alstom, την Philips, την Ευρωπαϊκή Εολική Ένωση και κάποιες άλλες τέτοιες επιχειρήσεις. Ε, είναι τιμή μου να βρίσκομαι εδώ πέρα σήμερα. Αυτό το οποίο λοιπόν θα ήθελα να σας πω είναι μια επιχειρηματική ιστορία για την ανάπτυξη και τις δουλειές στην Ευρώπη από μια εταιρεία αμερικανική αλλά με ε, σημαντική ευρωπαϊκή παρουσία στον τομέα αυτόν. Θα ήθελα να ξεκινήσω ε, κάνοντας βεβαίως την παρουσίασή μου. Αυτή είναι η παρουσία της General Electric στην Ευρώπη, στο χάρτη. Είμαστε εδώ πάνω από 100 χρόνια. Έχουμε 84.000 υπαλλήλους. Κάτι το ενδιαφέρον είναι όταν μιλάμε για καθαρές ε, τεχνολογίες. Ε, είναι πως δεν τα λέμε μόνο, αλλά τα κάνουμε και όλα σε αυτά που λέμε. Δηλαδή σε 7 χρόνια από σήμερα, το μάλλον τα τελευταία 7 χρόνια, από το 2004 μέχρι σήμερα αναπτύξαν πολλά πράσινα προϊόντα, μειώσαμε το αποτύπωμά μας κατά 1 τρίτο, ε, αυξήθηκε η ανακύκλωση του νερού κατά 30% και βεβαίω είχαμε και αύξηση των κερδών μας. Ε, δηλαδή είχαμε επενδύσει 5 δισεκατομμυρίων που δημιούργησαν έσοδα 20 δισεκατομμυρίων. Αυτό δηλαδή για να καταλάβετε πως ε, κατά την, ε, στο πλαίσιο της General Electric έχουμε τον πιο γρήγορα ψένομενο τομέα μας. Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη. Δύο παραδείγματα. Πρώτον, αιωλικά. Είμαστε αυτή τη στιγμή η κορυφαία εταιρεία στον κόσμο σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε χίλιους υπαλλήλους που απασχολούνται στην Ευρώπη μόνο στον τομέα των αιωλικών. Περιτώ να πω πως δεν βρισκόμαστε μόνο σε μερικά μέρη της Ευρώπης, βρισκόμαστε παντού. Αναπτύσσουμε παραδείγματο χάρη στη Ρουμανία, την το μεγαλύτερη εγκατάσταση αιωλικών ε, στην ξηρά στην Ευρώπη. Όλα αυτά δημιουργώντας θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Ένα άλλο παράδειγμα που είναι ενδιαφέρον γιατί δείχνει πόσο πολύ η δουλειά μας εδώ πέρα ε, εξάγεται εκτός Ευρώπης. Έχουμε μια πόλη ονομάτι Μπελφόρ, μπορεί να την ξέρετε. Εσείς ίσως έχετε πάει κιόλας. Μια μικρή πόλη στη Γαλλία. Μια περιοχή που έχει πληγεί από την αποβιομηχάνηση. Πήραμε από έναν ανταγωνιστή μια εγκατάσταση αιωλική, αλλά είχε ταυτόχρονα και αέριο και στροβίλους αερίου. Έχουμε λοιπόν γύρω στα 2.000 άτομα υπαλλήλους μας και οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται ε, με πλήρη απασχόληση εδώ στην Ευρώπη και το αντικείμενο τους είναι οι εξαγωγές. Είναι ανταγωνιστικοί. Οι πράσινες δουλειές αυτές ε, αφορούν τις εξαγωγές. 90% της παραγωγής του Μπελφόρ εξάγεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και 40% σχεδόν πάει σε χώρες Ασίας και Ειρηνικού και θα επανέλθω σε αυτή την περιοχή. Οπότε η πρωτοβουλία αυτή για τις χώρες ΑΠΕΚ σημαίνει ε, πώς θα έχετε νέες θέσεις εργασίας που θα κάνουν εξαγωγές στην εκλογική σας περιφέρεια. Και αυτό δεν είναι μόνο δικά μας νούμερα και σύμφωνα και με του υπολογισμού κομισιών ε, δεν είναι ψηλοπράγματα αυτά. Μιλάμε για 1.100.000 νέες θέσεις εργασίας ε, άμεσες και έμεσε στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και η ανάπτυξη αυτή, όπως είπα, ε, βρίσκεται τώρα στις αναδυόμενε αγορές. Το πρόβλημα είναι πω όταν πάμε να κάνουμε την εξαγωγή, για να εκμεταλλευτούμε αυτή την ανάπτυξη και να ξαναφέρουμε δουλειές στην Ευρώπη, αντιμετωπίζουμε προβλήματα εισόδου στην αγορά. Το πρώτο που αντιμετωπίζουμε είναι οι δασμοί. Οπότε δεν είναι σωστό να λέμε πως οι δασμοί στις καθαρές τεχνολογίες είναι ε, χαμηλοί. Είναι πολύ υψηλοί. Δείτε στην οθόνη. Ρωσία 10%, σε στροβίλους φυσικού αερίου, το Μεξικό 10% στις ανεμογεννήτριες ε, κτλ. Και όπως ανέφερε και ο Πίτερ Μπρούν από την ITCSD, είναι πώς ανταγωνιζόμαστε τα ορυκτά καύσιμα, τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας που δεν πληρώνουν δασμούς. Αυτές οι πηγές ενέργειας α, ε, θεωρούνται πρώτες ύλες και θέλουμε ίσως όρους ανταγωνισμού. Οπότε το να καταργήσουμε τους δασμούς είναι απολύτως απαραίτητο. Ο πράσινος προστατευτισμός, επίσης τα μη δασμολογικά εμπόδια, είδατε ήδη κάποιες διαφάνειες ε, για το πώς πολλαπλασιάζονται ε, οι διατάξεις για τοπική παραγωγή, για αντι-dumping, για τοπικό ποσοστό παραγωγής, για υποχρεωτική μεταφορά πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτά είναι τα πραγματικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές μας εξαγωγές για να α, πιάσουν αυτές τις αγορές. Και το αποτέλεσμα είναι πως σε κάποιες τέτοιες χώρες BRIC, παραδείγματο χάρη, το ποσοστό τη αγορά για τα αεολικά ήταν 70% πριν από 7 χρόνια, το, το δικό μα. Ε, είχε η Vestas, η General Electric, η Siemens και σε 7 χρόνια το ποσοστό των ευρωπαϊκών εταιριών έπεσε στο 10%. Δεν έγινε ε, ως διαμαγείας, ούτε αυτές οι χώρες ανακάλυψαν νέες τεχνολογίες. Είναι το αποτέλεσμα δασμών και μη δασμολογικών φραγμών. Και, ακόμη χειρότερο, έχουμε μια αγορά η οποία δεν είναι προβλέψιμη. Γιατί έχουμε πολλές διαμάχες ενώπιον του ΠΟΕ. Τα τελευταία δύο χρόνια είχαμε έξι νέες διαμάχες στον ΠΟΕ. Έχουμε λοιπόν απόδειξη του ότι υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την αγορά. Έχουμε εμπορικούς πολέμους. Πώς θα λυθεί αυτό. Μέσω ομινήσεων, εντάξει, είναι καλό για τους δικηγόρους. Ή με τις διαπραγματεύσεις. Και βεβαίως, ο πιο βιώσιμος τρόπος για να λύσουμε αυτά τα ζητήματα είναι να πείσουμε τις χώρες να επανέλθουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Τώρα, το αποτέλεσμα. Όλα αυτά σημαίνουν αυξανόμενο κίνδυνο, λιγότερη προβλεψιμότητα στον τομέα της καθαρής ενέργειας και όταν είσαι τραπεζίτης, όταν είσαι επενδυτικό ταμείο, αυτό το οποίο δεν σου αρέσει είναι ο κίνδυνος και η μη προβλεψιμότητα. Ποια είναι η συνέπεια? Έχουμε πτώση κατά 90% πέρσι των επενδύσεων στην καθαρή ενέργεια. Για πρώτη φορά είχαμε μεγάλη πτώση. Όπως βλέπετε και από την σχεδόν συνεχή αύξηση που είχαμε μέχρι τώρα. Βεβαίω υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, δεν είναι μόνο αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και το σχιστολιθικό αέριο, αλλά το περιβάλλον αυτό δημιουργεί μη προβλεψιμότητα και αβεβαιότητα. Οπότε αυτό το οποίο χρειαζόμαστε ειδικά σε καιρούς μείωσης της δημόσιας χρηματοδότησης είναι ίση ώρα ανταγωνισμού και να επιτρέψουμε στην παγκόσμια αγορά να αναπτυχθεί για να έχουμε μεγαλύτερη κλίμακα για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε έτσι, τις πιο παραδοσιακές πηγές ενέργειας. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, δεν θα σας προξενήσει η εκπλήξη, είναι μηδενικούς δασμούς, το να κατέβουμε στο 5% στις χώρες Ασίας, ε, Ασίας Ειρηνικού είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Πρέπει να κάνουμε αυτό το οποίο έκαναν και ε, άλλοι στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου υπήρχε η αίσθηση πως ξεκινούσε το διαδίκτυο οι εταιρείε υψηλή τεχνολογίας θα ήταν σε μια αγορά που θα άνθιζε, οι κυβερνήσεις συνεννοήθηκαν και είπαν πως η καλύτερη βοήθεια που μπορούσαν να δώσουν ήταν να ε, καταργήσουν τους δασμούς. Και κατέληξαν στη λεγόμενη Συμφωνία Περιπληροφορικής στον ΠΟΕ. Το ίδιο χρειαζόμαστε και εδώ. Είμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, αντιμετωπίζει κρίση αυτή τη στιγμή ο τομέα των ανανεώσιμων, χρειάζεται μια όθηση μέσω της κατάργησης των δασμών. Τι αποτέλεσμα θα έχει η κατάργηση των δασμών και των μη δασμολογικών φραγμών. Δεν αφορά μόνο εμάς στην General Electric, Αυτά τα στοιχεία που σας λέω είναι της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει υπολογίσει πως τα θετικά αποτελέσματα της κατάργησης δασμών και μη δασμολογικών φραγμών μπορεί να ανέλθουν σε μια αύξηση κατά 63% του μεγέθους της παγκόσμιας αγοράς για αυτές τις τεχνολογίες. Οπότε, πάλι μιλάμε για μια τεράστια όθηση. Πιθανές δράσεις. Έχουμε μια χρυσή ευκαιρία. Συμφωνούμε με αυτό το οποίο είπε η κυρία Σχαλτεμόζε για να κινητοποιηθούμε και να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία. Βεβαίως, ε, οι χώρες αυτές δεν είναι η, ε, το α και το ω. Και η συμφωνία αυτή δεν είναι τέλεια. Βεβαίως θα θέλαμε και άλλα προϊόντα να συμπεριληφθούν, αλλά είναι μία αρχή. Και είναι εύθραυστη αυτή τη στιγμή. Όπως είπαμε, συμφώνησαν σε αυτή τη συμφωνία γιατί είναι και μη δεσμευτική, οπότε το ερώτημα είναι Είμαστε διατεθειμένοι, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσουμε γνωρίζοντας πως το περιβάλλον αυτό και το εμπόριο αυτών των προϊόντων απασχολεί ευθύς εξ αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή θέλουμε να πούμε ε, δεν είναι τέλεια συμφωνία και δεν κάνουμε τίποτα τότε θα έχουμε την πολιτική ευθύνη για την αποτυχία ενώ είμαστε ε, πρώτοι στον κόσμο σε αυτές τις τεχνολογίες. Και αυτό δεν αφορά μόνο την μείωση των δασμών. Η συμφωνία αυτή μπορεί και να αφορά τα, ε, τους μη δασμολογικούς φραγμούς. Αν διαβάσετε την εντολή του ΑΠΕΚ και δεν είναι κάποιοι μυστήριοι διαπραγματευτές το κάνουν, έχει συμφωνηθεί στο επίπεδο του Πρόεδρου Ομπάμα, στο επίπεδο του ε, Πρωθυπουργού Σινχουά στην Κίνα και συμφώνησαν να υπάρξει και μεγαλύτερη διαφάνεια στις δημόσιες προμήθειες και που είναι ενδιαφέρον προδιαγραφές ρυθμιστικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο πρώτος εξαγωγέας αυτής της τεχνολογίας θέλει να παραμείνει εκτός αυτής της πρωτοβουλίας γνωρίζοντας πως η ε, περιοχή του ΑΠΕΚ ε, είναι αυτή τη στιγμή η πιο γρήγορα αναπτυσσόμενη ε, περιοχή στον πλανήτη κατά 5% σε ετήσια βάση. Οπότε έχουμε τα εξαγωγικά συμφέροντα της Ένωσης και το ενδιαφέρον είναι πως βλέπετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή τη στιγμή πρώτη στον κόσμο σε αυτό. Δεν είναι πως θα ανοίξει λοιπόν την πόρτα της ε, σε, σε φτηνά κινέζικα μπλουζάκια ας πούμε. Είναι πρώτη στον κόσμο στις 54 ε, καθαρές τεχνολογίες που ορίζει ο ΑΠΕΚ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη. Πρώτη την Γερμανία που θα επωφεληθούν από τη συμφωνία αυτή. Οπότε το μήνυμα είναι πως η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας οι δασμοί είναι ήδη κάτω από το 5%, χωρίς ένα κόστος, θα μεταμορφώσει μια τοπική περιφερειακή πρωτοβουλία σε κάτι το οποίο δυνητικά θα μπορούσε να είναι μια νέα συμφωνία του ΠΟΕ που σε τελική ανάλυση θα συνεισφέρει στην ενίσχυση του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Γιατί αυτό το οποίο θέλουμε όλοι σήμερα είναι να γίνει αυτή η συμφωνία και να ενταχθεί στον ΠΟΕ. Ο μόνος τρόπος για να γίνει αυτό είναι να ε, και να υπογράψει τη συμφωνία αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τρόπο για να μετατραπεί μια περιφερειακή μη δεσμευτική συμφωνία ε, σε μια συμφωνία του ΠΟΕ που θα ενισχύσει τον ΠΟΕ και θα επιτρέψει στι εταιρείε μα να ξαναφέρουν τις πράσινες δουλειέ και την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you all. Uh, moving to the second... Ευχαριστούμε. Περνάμε στο δεύτερο τμήμα αυτής της ακρόασης. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Μπορούν να έχουν τώρα το λόγο τα μέλη της Επιτροπής αυτής για να υποβάλουν ερωτήσεις. Κρίστοφα Φιέλνερ του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ πολλούς προβληματισμούς μπορεί να έχει κανείς, αλλά πρώτα απ' όλα μερικές απλές ερωτήσεις για τον πρώτο ομιλητή, τον κύριο Μπρεν, μας μίλησε για τοπικό περιεχόμενο και κάποιες διαφάνειες. Εγώ βρήκα κάποιες ε, Δεν είδα χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή τη διαφάνεια. Μπορείτε να μα το εξηγήσετε γιατί και όσον αφορά του εμπορικού περιορισμού ε, για τους ηλιακούς συλλέκτες. Υπήρχαν εκεί η Γαλλία και η Ιταλία. Ε. Θα ήθελα να ακούσω. Τι είναι αυτό. Ζητώ συγγνώμη για την έλλειψη των γνωσεών μου σε αυτό το τομέα, αλλά όσον αφορά την και ε, δεν είναι μόνο η ενέργεια κομμάτι των περιβαλλοντικών αγαθών. Ε, η λίστα ΑΠΕΚ συζητήσεται με την ενέργεια ως επιτοπλίστων, λιγότερο, γιατί ουσιαστικά αυτό μας ανησυχεί και μπορεί να είναι και πιο δύσκολο κομμάτι από άλλα πράγματα. Και ο διαχωρισμός, όπως έδειξε ο συνάδελφος της ΕΦΙΚ, μπορεί να είναι αρκετά περίπλοκος. Και μετά φυσικά όσον αφορά τη συμφωνία ΑΠΕΚ δεν είναι αυτή ε, συμφωνία καθαρής τεχνολογίας αλλά το θέμα είναι τι θα γίνει για παράδειγμα πιστεύω δεν μπορούμε εμείς να κάτσουμε στην άκρη και να πούμε αν ναι, συμφωνούν για μικρούς δασμούς ε, και το επόμενο που μπορεί να συμβεί είναι ότι θα υπάρξουν πραγματικά πρότυπα στα οποία εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε παρότι είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Αυτή είναι μια πτυχή που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είτε θα καθόμαστε στο τραπέζι να διαπραγματεύσουμε, είτε θα καθόμαστε και θα κοιτάζουμε τι κάνουν οι άλλοι. Πολύ ενδιαφέρον βρήκα τη μη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στη Γενέβη και κάτι άλλο περίεργο είναι ότι οι πράσινοι δεν βρίσκονται εδώ στην Επιτροπή αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται κάπως με όλο αυτό αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό το τομέα και εδώ δεν συμφωνώ με την ΣΕΦΙΚ αν έχουμε υψηλούς δασμούς σε έναν τομέα αυτό αποτελεί επιχείρημα να μην μειώσουμε τους δασμούς σε έναν άλλο τομέα γιατί αυτό είναι διακριτική μεταχείριση αν το εφαρμόσουμε αυτό τότε καλύτερα να διακόψουμε τις εργασίες της Επιτροπής γιατί τότε δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμένα αυτό που με ανησυχεί είναι αν εστιαστούμε μόνο στην ενέργεια την τελευταία φορά που έψαξα δεν βρήκα δασμούς για το πετρέλαιο, για το φυσικό αέριο ή για άλλα ορκητά καύσιμα. Το οποίο σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε στην εξή περίεργη κατάσταση. Όχι μόνο έχουμε δασμούς για ό,τι θέλουμε να προωθήσουμε, αλλά αυξάνουμε τους δασμούς αυτούς. Σε αυτή την επιτροπή μιλάμε για δασμούς αντι-dumping, είναι περίπλοκο γιατί έχει να κάνει και με άλλο θέματα, άλλες πτυχές της οικονομίας. Είναι σαν να λέμε ότι είναι σωστό, τι είναι λάθος, τέτοια πράγματα, αλλά είναι ενδιαφέρον ότι με τεράστια ακρίβεια καταφέραμε τώρα να έχουμε την αντι-dumping για όλους τους μορφές εναλλακτικών ενεργειών. Διοεθανόλη, ε, ηλιακούς συλλέκτες, ε, πολυσιλικόνες για ανεμογεννήτρες, όλα αυτά. Εάν αυτή δεν είναι η λύση, τότε ποια πρέπει να είναι η λύση. Για όλους όσου θεωρούν ότι αυτό είναι πρόβλημα. Σίγουρα θα ήταν καλύτερο να γίνει στο πλαίσιο του ΠΟΕ. Η ολοκλήρωση του γύρου της Ντόχα θα ήταν κάτι καταπληκτικό. Αλλά εγώ θα συνεχίσω να υπερασπίζομαι την ε, Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τις ΗΠΑ, για παράδειγμα. Και στο ίδιο πλαίσιο Εάν καταφέρουμε να συμφωνήσουμε κάτι, δεν είναι αυτό προτιμότερο από το να λέμε καταλαβαίνω την άψη του ΠΟΕ, αλλά δεν θα μας βοηθούσε αυτό, δεν θα σας βοηθούσε αυτό. Uh, Uh, next. Uh, That's good to hear. Χάσαμε το χρόνο μας με αυτά που είπατε. Πάλμερ της Γκουε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ενδιαφέρουσες αυτές οι συζητήσεις εδώ και Έχουμε μεγάλους οργανισμούς, μεγάλες εταιρείες όπως η General Electric, τις οποίες τα συμφέροντα φαίνεται να συμπίπτουν με τα συμφέροντα του περιβάλλοντος. Και υποτίθεται έχουμε μια ευχάριστη σύμπτωση μεταξύ των συμφερόντων των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος. Το ίδιο γίνεται όταν μιλάμε και για την ανάπτυξη, όπου πάλι συμπίπτουν τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων με το καλό του περιβάλλοντος από ιδεολογική άποψη κατά την απόψή μου, δεν συμπίπτουν. Δεν θα καθίσω τώρα να κρίνω την απελευθέρωση των περιβαλλοντικών αγαθών, αλλά πιστεύω ότι η ιδέα ότι δεν υπάρχει τριβή μεταξύ του καπιταλισμού, δηλαδή της κερδοσκοπίας και του περιβάλλοντος, ότι υπάρχουν, ότι μπορούν να συγκλίνουν, αυτό είναι λάθος. Μπορεί μια μεγάλη επιχείρηση να θελήσει να είναι μια εταιρεία καθαρή ενέργεια, αλλά είναι ένα από του μεγαλύτερου παράγοντε ρήπων στι Ηνωμένε Πολιτείε με επικίνδυνα υλικά. Ε, ρηπαίνει, έχει ρηπάνει το ποταμό σε μεγάλο βαθμό. Τώρα αυτά που μας λέει η GE λοιπόν ότι υποστηρίζει το περιβάλλον και ότι αυτό υποτίθεται είναι ωφέλιμο για τα κέρδη τους είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το εξετάσουμε ανεξάρτητα, με κάποια ανεξάρτητη αξιολόγηση. Αυτό που θέλω να πω ως γενικό σχόλιο είναι ότι ακόμη και αν η απελευθέρωση των περιβαλλοντικών αγαθών αποτελέσει αρρωγή, θα είναι ανεπαρκής αυτή η αρρωγή δεδομένη της κλίμακας της, κλίμακα, ε, της κρίσης που αντιμετωπίζουμε σε κλιματικά θέματα και δεν πρόκειται να αντισταθμίσει την απουσία σοβαρών δεσμευτικών στόχων και την απουσία προγραμματισμού. Έχω τρει ερωτήσει. Πρώτον, υπάρχουν μελέτε ανεξάρτητε σε σχέση με το ποιε είναι οι επιπτώσει και αυτή δεν η επιπτώσει πλήρους απελευθέρωση του εμπορίου περιβαλλοντικών αγαθών ή των 54 αγαθών που περιλαμβάνονται στο ΕΠΕΚ. Ποιε θα είναι οι επιπτώσει για τι εκπομπέ ε, αερίων θερμοκηπίου ή για άλλου πράγματα που αξιολογούμε όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Δεύτερον, πόσα από τα αγαθά που περιλαμβάνεται στη λίστα του ΑΙΠΑΚ ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, πόσα από αυτά ενδιαφέρουν τις χώρες, ε, τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι τα εξάγουν. Και τρίτον, όσον αφορά την υγεία και την περιβαλλοντική απόδοση και τη μέτρησή τους λαμβάνονται υπόψη η διαδικασίε και οι μέθοδοι όπω κάναμε και όταν συζητούσαμε για τα βιοκαύσιμα και όπω θα κάνουμε και για την αλλαγή χρήση γεών. Πώ αξιολογείται δηλαδή, το περιβαλλοντικό αγαθό και τι επιδόσει έχει. Καλά, εδώ δεν είναι, είναι τώρα διάλογος μόνο με την GE. Ε. ε. Θα μπορέσετε να απαντήσετε, φαντάζομαι, GE, σε αυτές τις ε, κατηγορίες. Ε, κύριε Γκασπάρη. Ευχαριστώ. Ε, είναι συναρπαστικά αυτά ε, που ακούμε για το τι διαφορετικές απόψεις έχει η βιομηχανία για αυτά τα πράγματα, αλλά αυτό το οποίο με ενδιαφέρει είναι αυτό το οποίο είπε ο εκπρόσωπος της χημικής βιομηχανίας. Είναι δηλαδή ε, δύσκολο να διακρίνουμε τι είναι περιβαλλοντικό αγαθό και τι όχι. Και άκουσα εγώ τον εκπρόσωπο της General Electric που είπε πως υπάρχει λίστα προϊόντων στις χώρες ε, Ασίας ε, Ειρηνικού που είναι περιβαλλοντικά αγαθά και ό,τι δεν είναι στη λίστα δεν θεωρείται περιβαλλοντικό αγαθό. Τι λέει λοιπόν στα επιχειρήματα του χημικού κλάδου πως δεν υπάρχει διαχωρισμός. Πώς κάνει το διαχωρισμό η General Electric. Τι είναι περιβαλλοντικό αγαθό και τι όχι. Γιατί είναι τελείως διαφορετική η περίπτωση αυτή από τη χημική βιομηχανία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέμπερ. Ο σου έλεγε ότι το δηλητήριο δεν βρίσκεται στην ουσία αλλά στη δόση. Αυτό περίπου μας είπε και ο εκπρόσωπος της χημικής βιομηχανίας ότι ένα προϊόν μπορεί να είναι εξαιρετικά χρήσιμο για κάποιες χρήσεις και ε, σε κάποια δόση, ενώ επιβλαβέστατο σε κάποιες άλλες. Και συμφωνώ με τον Πρόεδρο. Ο ορισμός αυτών των περιβαλλοντικών αγαθών είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή. Τι σημαίνει, από πότε ένα αγαθό είναι, μπορεί να θεωρηθεί ως ε, περιβαλλοντικό αγαθό ή περιβαλλοντική ζημία. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ένα άλλο θέμα που θέλω να θέσω είναι ότι μπορώ να αποδεχθώ ότι σήμερα πολλά προϊόντα είναι made in the world, γίνονται στον κόσμο κάπου αναφέρεται, δηλαδή στην Κίνα, αλλά η μείωση των τελωνιακών δασμών μπορεί να έχει μια κάποια λογική, αλλά ειδικά σε αυτό το τομέα και για την Κίνα αντιμετωπίζουμε ε, μαζικές ε, ε, δραστηριότητες dumping στον τομέα των φωτοβολταϊκών και των αιωλικών γεννητριών. Είμαστε πάρα πολύ μπροστά στην Ευρώπη και πάρα πολύ σχετικές βιομηχανίες γερμανικές καταστράφησαν από τη μαζική πλημμυρίδα προϊόντων παρεμφερών που προέρχονταν από την Κίνα με μεγάλες επιδοτήσεις, με εργασιακό κόστος μηδενικό, επιδοτήσεις από, τις, ε, από την κεντρική διοίκηση, από την περιφερειακή διοίκηση και αντιμετωπίζουμε και άλλου είδους κοινωνικά ντάμπ. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με όλες τις διαδικασίες αντι-dumping του ΠΟΕ και η μείωση, λαμβάνοντα όλα αυτά υπόψη, η μείωση των τελωνιακών δασμών είναι δευτερεύον θέμα. Τώρα, υπάρχει το θέμα της ε, μη ρύθμισης, δηλαδή της μη εφαρμογής κάποιων κανόνων και η καταπολέμηση όλων των μορφών dumping που θα ήθελα να μου εξηγήσουν ε, οι παρεμβαίνοντες. Ευχαριστώ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι τότε ας ακούσουμε και την Επιτροπή. Όχι, όχι, η Κριστιάνα Μοσκαρντίνη, δίπλα μου, δεν σε είδα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, απλά να πω ότι συμφωνώ με τις παρεμβάσεις των συναδελφών. Πιστεύω ότι πρέπει να έχει προτεραιότητα μια οριστική διαφάνεια όσον αφορά τα συστήματα συμπεριφοράς, διότι πολλές φορές συναντάμε διαφορετικές απαντήσεις ανάλογα με το θέμα και τα προβλήματα του anti-dumping, των διαδικασιών dumping, τα προβλήματα της Γερμανίας και τα προβλήματα της Ιταλίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε αυτόν τον τομέα είναι τρομακτικά. Πριν προχωρήσουμε λοιπόν παραπέρα, χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες και βεβαιότητες, διότι η Ευρώπη δεν μπορεί να συνεχίσει να ακολουθεί αυτή τη διαδικασία χωρίς να λαμβάνει κανένα αντάλλαγμα. Ευχαριστώ. Ωραία, λοιπόν, ας ακούσουμε τώρα στην Κομισιόν, κυρία Χένξε. Ευχαριστώ πολύ που μου δίδετε το λόγο. Και θα σχολιάσω μετά από τις συγγύσεις των ομιλητών και τις ερωτήσεις που έγιναν. Θα ήθελα να τονίσω ότι στην Επιτροπή υποστηρίζουμε πάρα πολύ την χρησιμοποίηση όλων των μέσων που διαθέτουμε για την απελευθέρωση των περιβαλλοντών αγαθών και υπηρεσιών. Βεβαίως, η πολυμερής απελευθέρωση είναι το ευκταίο. Ανέφερε η κυρία Μότα τι έγινε σε επίπεδο γύρου της Ντόχα για την απελευθέρωση αυτών των προϊόντων. Δέκα χρόνια κρατούν οι διαπραγματεύσεις, αλλά στην ιστορία δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα προβλήματα υπάρχουν. Πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Πρώτα απ' όλα έλλειψη δεσμεύσεων και από τις ε, αναπτυγμένες και από τις ε, αναδυόμενες ε, χώρες. Και χαίρομαι που άκουσα κάποια σχόλια εκ μέρους της ADCT που ανέφερε αυτό το θέμα. Δεύτερο πρόβλημα, και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο ανέφερε και το ΣΕΦΙ και η χημική βιομηχανία, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσει κανείς να συμφωνήσει για το τι είναι ε, καθαρά αγαθά και πράσινα. Ο ρεαλισμός και ο πραγματισμός είναι κάτι το οποίο ανέφερε και στην άλλη του Νομίζω ότι αυτό που έκανα δεν ήταν ε, ακαδημαϊκές συζητήσεις, αλλά παρέθεσαν ένα κατάλογο περιβαλλοντικών αγαθών. Και ίσως θα πρέπει να σχολιάσω για κάποια από τα αγαθά που περιλαμβάνω στον κατάλογο αυτό. Μιλούμε για ομάδες ε, ε, ανανεώσιμων ε, πηγών ενέργειας, για νέες καθαρές τεχνολογίες. Πρόκειται κυρίως για αγαθά τα οποία είναι φιλικά προς το περιβάλλον, και καθαρά προϊόντα. Παρά το για όλα δεν έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη. Και βεβαίω οι συζητήσεις δεν έγιναν συζητήσεις και για τα μη τελωνιακά, μη, μη τελωνιακούς θασμούς Πριν από ένα χρόνο έγινε και συζήτηση για τα NTB, για τους μη δασμολογικούς φραγμούς. Και αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Βλέπουμε ότι στη Γενέβη υπάρχει νέος πρόεδρος στην σχετική επιτροπή, θέλει να συνεχθεί ο διάλογος, εμείς συνεχίζουμε και συνεχίζεται η εξερεύνηση και άλλων διάβλων. Θέλουμε επίσης να δούμε Επίσης, πώς θα μπορέσουμε κάτι που δεν έγινε στο παρελθόν να εκμεταλλευτούμε το γεγονός της κριτικής μάζας, διότι όπως καταλαβαίνετε η Κίνα είναι μέρος αυτής. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι έτσι ως έχει η πρωτοβουλία, η ΠΑΚ, δεν θα προσχωρήσουμε την εμείς. Σας θέλω να σας καθησυχάσω. Χαιρετίζουμε σε αυτή την πρωτοβουλία και θα πρέπει να, δούμε, να παραδεχθούμε ότι πρόκειται για μια, ένα πρώτο κατάλογο προϊόντων στα οποία συμμετέχουν τόσε χώρε. Θα πρέπει να δώσουμε χρόνο στην ΕΠΑ ώστε να μπορέσει να παγιώσει και να οριμάσει αν θέλετε αυτή την πρωτοβουλία. Δεν είναι δεσμευτική υπό τους όρους της ΠΟΕ, δεν υπάρχει θέμα διεφυλικές προ το καρόν, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον και Περιμένουμε ότι όλοι οι εταίροι μας θα συζητήσουν αυτό το θέμα στα πλαίσια των ε, ε, εξελίξεων των συζητήσεων στη Γενευκή θα υπάρχει και μία νέα πρωτοβουλία IPAC+. Πρόκειται λοιπόν για εναλλακτικέ ενδεχομένω λύσεις για το μέλλον. Και βεβαίως ίσως και εκείνους θα τους ενδιαφέρει να προσχωρήσει στην πρωτοβουλία αυτή και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα, από την ε, ευρωπαϊκή προοπτική, τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την πρόσβαση στην αγορά. Η πρωτοβουλία ή θα σημαίνει εφικτά ωφέλη. 54 αγαθά είναι ένα μικρό ποσοστό στα πλαίσια του εμπορίου, αλλά ο, κυρίως εξαγωγές τέτοιων αγαθών είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για ένα τομέα που εξελίσσεται. Οι εξαγωγέ έχουν αυτά τα δύο τελευταία χρόνια κατά 10%. Το 60% πηγαίνουν προ τι χώρε ΙΠΕΚ και το 1 τρίτο ή να μην πω το 50% πηγαίνουν στι χώρε ΙΠΕΚ που έχουν του υψηλότερο επίπεδο ε, δασμών. Σε αυτή την κατάσταση λοιπόν κρίση, νομίζω ότι αυτή η δυνατότητα είναι ενδιαφέρουσα και θα δούμε εάν θα γίνει κάτι στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και συζητήσεων σε επίπεδο ΠΟΕ στη Γενέβα. Από πλευράς περιβάλλοντος. Σύντομα θα πω ότι πρόκειται για έναν περιβαλλοντικά υγιή κατάλογο αγαθών. Θα υπάρξουν ωφέλη για το περιβάλλον και από πολιτικής ε, πλευράς η Ευρώπη θέλει να έχει τον ηγετικό ρόλο. Τελευταία και αλλά όχι λιγότερο σημαντικά πρέπει να σας πω ότι τα απελευθέρωση των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών είναι κάτι το οποίο και εμείς προωθούμε σε επίπεδο FDA. Θέλουμε να υπάρξει απελευθέρωση ε, με κάποιες χώρες χωρίς μεταβατικές περίοδους, στην Σιγκαπούρη, στην Κορέα, στην Κολομβία και άλλες χώρες. Επίσης έχουμε συμπεριλάβει εδώ νέα ε, κεφάλαια για αγαθά και υπηρεσίες πράσινες και υπάρχει και μία καινοτόμος προσέγγιση με χώρες νοτιοαλλατικής Ασίας που αφορούν ε, μη, δασμ, μη, ε, δασμολογι, τελωνιακούς δασμούς και μη δασμολογικούς φραγμούς σε θέματα ενεργειακά. Αναφέρθηκαν επίσης ε, διάφορα για τις δασμολογικούς και μη δασμολογικούς φραγμούς. Νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε μία ολιστική ε, ε, προσέγγιση του όλου θέματος. Θα πρέπει να δούμε το θέμα της επίλυσης, των μηχανισμών επίλυσης διαφορών, πώς θα διαμορφωθεί και νομίζω ότι θα πρέπει ούτως ένα στον τομέα αυτό όλοι να βρίσκονται σε ίδια βάση. Τελειώνοντας, θα θέλω να πω ότι θα συνεχίσουμε σε όλα αυτά τα μέτωπα, διμερός, πολυμερός και σε όλα τα επίπεδα, γιατί πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα θέμα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι η επιπτώσεις για το εμπόριο αυτών των θεμάτων που αφορούν τα περιβαλλοντικά αγαθά και υπηρεσίε, είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πρόκειται για μια νέα, λοιπόν, για μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική, την οποία δεν θέλουμε να σημασία δεν θέλουμε να παραγνωρίσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Τρίτο μέρος αυτής της ακρόασης ακούσουμε ξανά τους προσκεκλημένους μας ώστε να απαντήσουν στις ερωτήσεις. και στις επιφυλάξεις που εξέφρασαν τα μέλη της Επιτροπής συμπεριλαμβανομένου φυσικά και του ζητήματος του ορισμού, κατά πόσο υπάρχει ορισμός των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών. Κατά πόσο η συμφωνία είναι κάτι που θα πρέπει να γιορτάσουμε ή αν δεν έχει καθόλου νόημα ή αν θα αποτελέσει το επόμενο βήμα για να προωθήσουμε την πρωτοβουλία τη Κομισιόν σε αυτόν τον τομέα. Λοιπόν, θα ακολουθήσω την αντίστροφη σειρά των ομιλητών. Ο πρώτος μας ομιλητής αυτή τη φορά θα είναι ο κ. Φαμπιάν Ντελκρό. Και φυσικά έχετε την ευκαιρία, εφόσον το επιθυμείτε κ. Ντελκρό, να απαντήστε στις ε, κατηγορίες κατά της G. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ όλους για τις πολύ καλές αυτές ερωτήσεις. Ουσιαστικά η πρώτη ερώτηση αφορά τον ορισμό, η δεύτερη αφορά το κατά πόσο η G είναι κακιά και το, η τρίτη ερώτηση αφορά το dumping ουσιαστικά. Θα τις πάρουμε τη σειρά. Όσον αφορά τον ορισμό, συμφωνώ σε μεγάλο βαθμό με την έκκληση της Κομισιόν για ρεαλισμό. Οι χώρες εδώ και πάνω από 10 χρόνια στο πλαίσιο του ΠΟΕ προσπαθούν να, να συμφωνήσουν σε ένα θερισμένο ορισμό. Είναι ενδιαφέρον από ακαδημαϊκή άποψη και έχω μεγάλο σοβασμό προς τους ακαδημαϊκούς, αλλά δυστυχώς δεν έχει αποφέρει καρπούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας μια λίστα ατελή και τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο αξίζει να υπάρχει και τι θέλουμε να κάνουμε με αυτή, αν θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να μετατράπει σε κάτι δεσμευτικό, σε ένα ορόσημο ή κατά πόσο ενδεχομένω δεν θα καταφέρουμε να δράξουμε αυτή την ευκαιρία. Αυτός είναι, αυτό το μεγάλο ερωτηματικό σε σχέση με αυτόν τον ορισμό. Ενδεχομένως ε, αυτό που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θεωρεί ότι πρέπει να βελτιωθεί αυτή η λίστα, θα μπορούσε να συμπεριλάβει σε αυτήν καινοτόμες ιδέες όπως ε, να προτείνει στην ΕΠΕΚ να υιοθετήσει ένα μηχανισμό ενημέρωση τη λίστα, τακτική ενημέρωση διότι εν σε τελική ανάλυση δεν πρόκειται να σταματήσει η τεχνολογία, θα συνεχίσουν νέες ε, εφευρέσεις και από την κακή General Electric. Δεν βλέπω λοιπόν για ποιο λόγο δεν θα μπορούσαν να προσθεθούν εν τέλει χημικά προϊόντα σε αυτή τη λίστα. Φυσικά χημικά προϊόντα υπάρχουν τα οποία βοηθούν στην, στον καθαρισμό του νερού που περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα και εν τέλει η χημική βιομηχανία θα επωφεληθεί από μια πιο ελεύθερη αγορά. Τώρα κατά πόσο η General Electric είναι μεγάλη και σατανική και αν ε, βλάπτει το περιβάλλον. Τα πράγματα δεν είναι ούτε άσπρα ούτε μαύρα. Αν ρωτήσουμε τους ενα ε, εκατομμύριο ανθρώπους που υποστηρίζουν τις πράσινες επιχειρήσεις και τους πούμε ότι τους ρωτήσουμε κατά πόσο η G δεν συμβάλλει στην πράσινη ανάπτυξη θα έλεγαν ότι αυτό είναι λίγο αφηρημένο. Είναι μεγάλη εταιρεία, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι κακή. Αλλά εν τέλει εμείς καλούμαστε να ανταγωνιστούμε με κρατικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν μεγάλες επιδοτήσεις από τα εθνικά κονδύλια και ξέρετε τι, το να είναι μια εταιρεία μεγάλη αυτό της δίνει ευκαιρίες, μπορεί να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια αμερικάνικα δολάρια μέχρι το 2015 σε καθαρές τεχνολογίες. Αυτό είναι σημαντικό σε σχέση με τους μερικούς δημοσιονομικούς περιορισμούς. Φυσικά καμία επιχείρηση δεν είναι τέλεια. Και εμείς μαθαίνουμε από τα λάθη μας και το κάνουμε με μεγάλη χαρά. Το τρίτο σημείο που αφορά το dumping είναι πώς θα μπορούσε να προστατευτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, να συνεχίσει να προστατεύεται από αρπακτικές πρακτικές. Είναι μήπως σωστή στιγμή να στείλουμε ένα μήνυμα που θα πούμε ότι μονομερός θα προχωρήσουμε σε παροπλισμό η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δασμό 1,8% στη λίστα της ΑΠΕΚ. Αυτή, αυτός είναι ο επωνομαζόμενος προστατευτισμός που έχουμε, 1,8%. Κανένας σε αυτή την αίθουσα δεν θα πιστέψει ότι ένας δασμός του 1,8% αποτελεί προστατευτικό μέτρο. Είναι μια τιμή που θα μπορούσε να πληρώσει κανείς για να μπει στην αγορά ΑΠΕΚ. Έτσι θα πρέπει να το δούμε και μια πιθανή συμφωνία για την ελευθέρωση των καθαρών τεχνολογιών θα, μια τέτοια συμφωνία θα μας εμποδίσει καθιονδήποτε τρόπο από το να προστατέψουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν ε, υιοθετήσουμε συμφωνία με την ΑΠΕΚ θα εγκαταλείψουμε τους δικούς μας μηχανισμούς όχι θα συνεχίσουμε να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ε, στο πλαίσιο του ΠΟΕ και για το αντι-dumping και όλες τις σχετικές συμφωνίες. Αντιθέτως λοιπόν μάλιστα δεν πρόκειται να χάσετε τίποτα όσον αφορά προστατευτικά μέτρα και εργαλεία εκτακτής ανάγκης όπως χρησιμοποιούν όλα τα μέλη του ΠΟΕ αλλά ταυτόχρονα θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στον τομέα των εξαγωγών περιβαλλοντικών αγαθών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ακολουθεί ο κ. Ρενέ Σλότεν από την ΣΕΦΙΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα για το ερώτημα που αφορά την αύξηση των δασμών. Εγώ δεν είπα πως ήμουν υπέρ. Αντιθέτως, ε, είπα πως αν ε, είναι να βάλουμε στους δασμούς περιβαλλοντικά κριτήρια, ηθικά κριτήρια και δώσουμε προβάδισμα σε κάποια αγαθά, τότε οι υπόλοιποι δασμοί πρέπει να διατηρηθούν. Αυτό λέτε. Ε, εγώ δεν είπα αυτό το πράγμα, αντιθέτω. Θέλω απλά να επισημάνω πως δεν είναι πολύ λογική η όλη προσέγγιση. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω πως ήμουν σαφής ε, όσον αφορά τα ζητήματα του ορισμού. Δεν θα επανέλθω. Θα ήθελα να πω λίγα λόγια για το dumping ε, που γίνεται. Γιατί η χημική βιομηχανία έχει ξεκάθαρο ότι θέμα. ελεύθερο εμπόριο. Πρέπει να καταργηθούν όλοι οι δασμοί. Θέλουμε ελεύθερο εμπόριο. Αλλά και δίκαιο εμπόριο. Και θέλουμε σωστά μέσα προστασίας απέναντι στον αθέμητο ανταγωνισμό. Και μια που είμαι στην Επιτροπή σας θα ζητήσω ή ο εξυγχρονισμός ε, των ε, πολυμερών δεσμολογικών ε, συμφωνιών δεν θα πρέπει να εξασθενήσει την προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειαζόμαστε και δίκαιο εμπόριο. Δίκαιο εμπόριο μπορεί να υπάρξει μόνο όταν έχουμε και σωστά μέσα κατά του άδικου, αθέμητο ανταγωνισμό. Όσον αφορά λοιπόν τώρα την απελευθέρωση του, του θέματος, αυτό το οποίο χρειάζεται θα έλεγα ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι μια ευρύτερη μείωση των δασμών, όχι στοχευμένη και βασικό έργο του ΠΟΕ είναι η απελευθέρωση του εμπορίου και νέοι κανόνες όπως αναφέρθηκε και από τον κύριο Αμπτελ Μουτάλ. Και ο αυτή τη στιγμή δεν ε, έχει κάποια αποτελέσματα. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή μια φιλόδοξη συμφωνία ανάμα με κάποιους τομείς και μετά να προσθέσουμε και κάποιους, ε, κάποια περιβαλλοντικά αγαθά. Αυτό είναι το θέμα, όχι μόνο ένας κλάδος περιορισμένος, Ευχαριστώ κυρία Αμπτελμουτάλ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας σε κάποια ερωτήματα που ε, υπήρχαν αν θέλετε στα σχόλια του συναδέλφου από τη χημική βιομηχανία και μετά σε κάποια από τα ερωτήματα των βουλευτών. Κοιτάξτε, εγώ ασχολούμαι με αυτές τις διαπραγματεύσεις στον πω, εδώ και 10 χρόνια και ε, θεωρούσα πως μέχρι τώρα είχα ακούσει ε, οποιαδήποτε πιθανή αντίρρηση. Αλλά πρέπει να ομολογήσω πως οι αντιρρησει που γύρατε είναι καινούργιες για μένα. Είπατε πως θα έχουμε έτσι διακριτική μεταχείριση των προϊόντων που είναι εκτός λίστας. Εμείς λέμε πως πρέπει, πρέπει να διακρίνουμε μεταξύ ε, παραγόντων παραγωγή και τελικού προϊόντο. Δεν τα έχω ακούσει ποτέ αυτά τα επιχειρήματα εδώ και 10 χρόνια και μου προξενεί εντύπωση. Ο λόγο για τον οποίο χρειάστηκαν 10 χρόνια αυτέ τι διαπραγματεύσει είναι το ότι υπάρχει διαφωνία όσον αφορά το επίπεδο φιλοδοξία. Δεν έχω ακούσει ποτέ καμία χώρα του ΠΟΕ τα τελευταία 10 χρόνια να λέει πω ε, δεν χρειάζονταν ε, διαπραγματεύσει. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό, υπήρξαν κάποιε ερωτήσει για το εάν ε, η λίστα του ΑΠΕΚ αφορά μόνο ε, προϊόντα ενέργειας. Να απαντήσω. Η λίστα περιλαμβάνει έλεγχο, ε, εξοπλισμό ελέγχου της ε, ε του αέρα, προϊόντα ΑΠΕ, προϊόντα διαχείρισης αποβλήτων και λιμάτων, οπότε δεν είναι μόνο ενεργειακά προϊόντα. Επίσης έγινε ένα ερώτημα για το εάν έχει υπάρξει κάποια μελέτη για το τι θα σημάνει η απελευθέρωση και των 400 αυτών προϊόντων. Ε, είναι αδύνατο να γίνει μια τέτοια μελέτη γιατί η απελευθέρωση του εμπορίου δεν σημαίνει πω μια χώρα θα αρχίσει να το εισάγει την επόμενη μέρα. Εγώ είμαι Αιγύπτια και μπορώ να σα πω πω η χώρα μου δεν έχει πολλού περιβαλλοντικού κανόνε. οπότε το να φύγει ο δασμό στου καταλήτες δεν σημαίνει πω οι Αιγύπτιοι θα αρχίσουν αμέσω να εισάγουν περισσότερου καταλήτε γιατί δεν υπάρχει ανάλογη περιβαλλοντική νομοθεσία που να το απαιτεί. Οπότε υπάρχουν πολλά ε, ζητήματα που θα πρέπει να επιληθούν για να αντιμετωπίσουμε ε, αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, οι δασμοί είναι μόνο ένα από τα βήματα σε μια μακρά πορεία. Μία ερώτηση έγινε για το εάν ε, εξάγουν αναψώμενες χώρες τα προϊόντα αυτά. Ναι, βεβαίω. Κάποιε αναπτυσσόμενε χώρε είναι στην ε, πρωτοπορία και κάνουν πολλέ εξαγωγέ τέτοιε. Κίνα, Νότια Κορέα, Μαλαισία, Ινδονησία. Και πολλέ είναι και στην πρωτοπορία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνία τη τεχνολογία και ο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός ιδιοκτησία Ιδιοκτησίας έχει τα νούμερα που το επιβεβαιώνουν οπότε δεν εξάγουν απλά αλλά παράγουν την καινοτομία. Ο ίδιος κύριος είχε ε, ρωτήσει το εάν υπάρχει κάποια ε, διάκριση μεθόδων ε, παραγωγής και επεξεργασίας. Όχι, είναι πολύ πολύπλοκη αυτή η διάκριση και αποφάσισαν οι χώρε ότι καλύτερο είναι να μην γίνει κάτι τέτοιο. Απλά θα αναφέρουν τα προϊόντα χωρίς να ανοίξουν το δύσκολο αυτό κεφάλαιο που μετά δεν θα κλείνει. Άλλη μία ερώτηση ήταν το μήπως ο κατάλογος αυτός θα μπορούσε να διευκολύνει μια συμφωνία στον ΠΟΕ και αν ο ΠΟΕ είναι ανοιχτό σε ε, πρωτοβουλίες που γίνονται αλλού. Πράγματι εμείς θέλουμε να αποτελέσει ένα ορόσημο και εμείς το θεωρούμε κάτι το θετικό και όχι μία απειλή και μάλιστα όσον αφορά τη συμφωνία ελευθερίου εμπορίου, ο είναι ανοιχτό. αρκεί να δημιουργούν περισσότερο εμπόριο. Οπότε δεν έχουμε πρόβλημα με την λίστα αυτή. Ε, αντιθέτως θέλουμε να επεκταθεί. Τώρα κάποιες ερωτήσεις που είτε αναφέρουν άμεσα το ζήτημα του ντάμπινγκ, την επιδότηση των εξαγωγών από τις άλλες χώρες, άλλες χώρες ε, επιδοτούν τις εξαγωγές τους και μήπως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα βλάψει αυτόν με το να μειώσει τους δασμούς και γιατί η Ευρώπη να προσφέρει κάτι χωρίς αντάλλαγμα. Συνδέονται αυτά. Η απάντησή μου είναι πως βεβαίως το dumping είναι μια κακή πρακτική, αλλά δεν νομίζω πως ε, για να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα άλλο, το dumping θα το αντιμετωπίσουμε αντιμετωπίζοντα το dumping, όχι με δασμού. Και αυτό πρέπει να γίνει μέσω μια συμφωνία του ΠΟΕ για τι επιδοτήσει και τα αντίμετρα με τα μέσα που έχει ο ΠΟΕ και πρέπει να ενισχυθούν αυτά τα μέσα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μια σχετική διαπραγμάτευση, αλλά δεν νομίζω πως σωστή απάντηση είναι να δημιουργηθεί ένα άλλο εμπορικό πρόβλημα που πάλι τριβέ θα δημιουργήσει. Όσον αφορά το ότι δίνετε κάτι χωρί αντάλλαγμα. Η έκκλησή μου στην Επιτροπή σας είναι να θυμάστε πως πρόκειται για περιβαλλοντική διαπραγμάτευση. Αυτό το οποίο δίνει η Ευρώπη δεν σημαίνει πως θα το λάβει ως αντάλλαγμα ε, με βάση εμπορικές ε, παραχωρήσεις. Αυτό το οποίο θα λάβει το αντάλλαγμα είναι καλύτερο περιβάλλον. Οπότε, εάν... Οπότε, ε, όταν οι άλλοι θα χρησιμοποιούν περισσότερους καταλύτες, ε, περισσότερο εξοπλισμό διαχείρισης ε, αποβλήτων, λιμάτων κτλ. Η Ευρώπη κερδίζει ως προς το πιο καθαρό περιβάλλον. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ και για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της συζήτησης ο κύριος Πίτερ Μπρούν ICTS από τη Γενέβη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφέρω και το θέμα του πεδίου εφαρμογή. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι το πολυμερές σύστημα και ο γύρος της ΔΟΧΑ βρίσκονται μπλοκαρισμένα. Όλοι θέλουμε να περάσουμε στον επόμενο γύρο το συντομότερο δυνατό, αλλά υπάρχουν πολύπλοκα προβλήματα. Θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να καταλήξουμε στον στόχο που θέλουμε να υλοποιήσουμε και θα πρέπει να δούμε τα πράγματα με νέο, ρίχνοντας ένα νέο φως πάνω στο όλο αυτό το θέμα, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις για τις συμφωνίες με την περιβαλλοντική διάσταση. Εάν θέλουμε να έχουμε ευθύ εξ αρχής έναν ε, ιδεατό κατάλογο με όλα τα προϊόντα, ίσως αυτή να ήταν ε, μία πρώτη φιλοδοξία. Είναι διαφορετικό ε, τα πράγματα σήμερα, διότι ευθύ εξ αρχής είχαμε να κάνουμε με λίγες αρχές, με έναν πολύ δίσκαμπτο ε, κατάλογο το 96, αλλά τότε τι έγινε. Ε, επινοήθηκε ο μηχανισμός που είπαμε πώς θα πρέπει να εφαρμοστεί. Και είδαμε τι έγινε. Πρόκειται για μία προσέγγιση επιτυχή που δεν δημιουργεί πρόβλημα στους ε, στον γύρο διαπραγματεύσεων. Το θέμα είναι, μπορούμε να επαναλάβουμε τώρα το ίδιο μηχανισμό. Θα πω στους ε, φίλους της ΕΠΙΚ, το καλύτερο είναι ο εχθρός του κακού, όπως λέμε. Υπάρχει συνεκτικότητα ε, όσον αφορά κάποιους ε, δασμούς και μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχει συνεκτικότητα, σύγκληση απόψεων, συμφωνία ή κάποιον, αλλά δεν θα πρέπει ε, πάντα να ψάχνουμε πάντα το καλύτερο. Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι ο καλύτερος μηχανισμός που να εφαρμόσουμε και ας προχωρήσουμε. για να μπορέσει να τεθεί σε εφαρμή το σύστημα θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις και να το αφήσουμε να λειτουργήσει και θα δούμε μετά. Θα δείξει το μέλλον τι έχουμε κάνει. Ναι, στην ε, τελευταία χρονιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε δει να υπάρχει και διαφοροποίηση και εξελίξεις ανάλογα με, τον, ε, με τους διάφορους ε, τομείς. Ηλιακή ενέργεια, να αναφερθούμε στην ενέργεια ή με τις ανεμογεννήτριες. Και έχουμε δει ποιες είναι οι εξελίξεις. Και επίσης να διευκρινίσω το εξής. Η υπόδειξή μας δεν είναι να αλλάξουμε τους κανόνες ε, για στον ΠΟΕ για τους, ε, που πρέπει να ισχύουν για το εμπόριο. Απλώς θέλω να επαναλάβω ότι εδώ διακυβεύονται πολλά συμφέροντα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια πολλά υποσχόμενη βιομηχανία. Τα πράγματα αλλάζουν και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προχωρήσει εάν θέλει να, είναι, να έχει τον ηγετικό ρόλο ε, μία πολιτική φιλόδοξη. Οι τάσεις διαγράφονται και δεν μας περιμένουν εμάς για να καθοριστούν. Εμείς πρέπει να δούμε ποιες είναι οι τάσεις και να προλάβουμε κάποια γεγονότα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Ε, κάποια τελική παρατήρηση της Κομισιόν επί του θέματος. Ήθελα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να αναφέρω ότι μια της πρότασης που έκανα έκαναμε στην τελευταία Επιτροπή Εμπορίου και Περιβάλλοντος στη Γενέβη για το πώς να προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις, στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, ήταν μια ημερίδα με τη βιομηχανία για να μάθουμε τις νέες τάσεις όσον αφορά τα πρότυπα τεχνικών απαιτήσεων, τις υπηρεσίες μη δασμολογικών φραγμών και, κάναμε μια... και μετά να κάνουμε μια πρόταση στη γραμματεία για το πώς θα προχωρήσουμε και ελπίζω να συμμετέχει η βιομηχανία σε αυτό. Αυτή η τεχνική εργασία θα στρώσει το έδαφος ώστε η πρωτοβουλία αυτή να περάσει στο ΠΟΕ αυτό χρειάζεται να κάνει η να προωθήσει την εργασία αυτή. Ο συνάδελφο από την είπε ότι ο ορίζοντας βιομηχανία είναι δύο χρόνια και όχι δέκα. Θα ήθελα επίση να αναφέρω ότι η Κίνα θα φιλοξενήσει το ΕΠΑΚ το 2014. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Η Κίνα θα αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να προωθήσει την πρωτοβουλία αυτή. Σίγουρα τη συμφέρει να δεσμευτεί για την απελευθέρωση και πιστεύω ότι το 2014 θα αποτελέσει κρίσιμη χρονιά για αυτό το θέμα. Ε, thank you very much for... Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την άριστη, εξαιρετική ακρόαση. Πιστεύω ότι ήταν σωστή πρωτοβουλία για μια τέτοια ακρόαση και έγκαιρη, επίκαιρη. Είχε απόλυτο νόημα να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλο εξαγωγή σε αυτόν τον τομέα, γι' αυτό πρέπει να υποστηρίξουμε την απελευθέρωση αυτού του τομέα. Πόσο μάλλον επειδή οι περισσότεροι εμπορικοί μα εταίροι έχουν πολύ υψηλού δασμού σε αυτόν τον τομέα. Η συμφωνία ΕΠΕΚ ε, ενώ είναι πολύ περιορισμένη και μη δεσμευτική παραμένει θετική ρηξικέλευθο πρωτοβουλία και δεν πρέπει να αμελούμε τις επιπτώσεις της, τις συνέπειές της, είναι κάτι πάνω στο οποίο πρέπει να οικοδομήσουμε, να το χρησιμοποιήσουμε ως βάση και να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία ΕΠΕΚ συν, όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να σας υπενθυμίσω ότι ένας από τους στόχους της στρατηγικής 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πράσινη ανάπτυξη και συνταγματικά και πολιτικά έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε βάσει μιας φιλοσοφίας ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Θα μου έκανε λοιπόν έκπληξη να μην υποστηρίξει η Κομισιόν την ιδέα της απελευθέρωσης των περιβαλλοντικών αγαθών και υπηρεσιών στο πλαίσιο συμφωνίας. Και όπως είπε και ο τελευταίο ομιλητής, ο κ. Μπρούν, πολύ σοφά και χρησιμοποιώντας επιχειρήματα, ο πρόεδρος της ITA ε, το είπε ότι οι συμφωνίες αυτές δεν είναι σύμβατες με τους κανόνες του ΠΟΕ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με χαμηλές προσδοκίες πάνω στις οποίες θα οικοδομήσουμε ώστε να καταλήξουμε σε μια πολύ φιλόδοξη συμφωνία. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους συμμετείχαν σε αυτή τη συζήτηση, τους συναδέλφους μου αυτής της Επιτροπής, τη Γραμματεία που οργάνωσε αυτή την ακρόαση, τους ομιλητές μας. Είστε ευπρόσδεκτοι στο κοινοβουλίο μας, είμαστε πάρα πολύ ανοιχτόμυαλοι και πάντα είμαστε διατεθειμένοι να ακούσουμε τους προσκεκλήμενους μα και φυσικά, όπως πάντα, την Κομισιόν που συμμετείχε δραστήρια στη συζήτησή μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερως. And, uh, our next item is... Το επόμενο σημείο μας είναι το σημείο 15. Which will uh, be an exchange of views with ανταλλαγή ε, απόψεων με τον Επίτροπο Ντεχούχτ, ο οποίος ε, θα βρίσκεται μαζί μας σε μερικά λεπτά. Ας αφήσουμε λοιπόν τους προσκεκλημένους, ας αφήσουμε το χρόνο στους προσκεκλημένους μας να αποχωρήσουν. Εφόσον το επιθυμούν φυσικά αλλιώς μπορούν να καθίσουν και να ακούσουν τον κύριο Επίτροπο. μέχρι να φτάσει ο κύριος Επίτροπος ε, ας κάνουμε ένα πεντάλεπτο διάλειμμα. May I have attention, please? Uh, την προσοχή σας παρακαλώ. Συνεχίζονται οι εργασίες με την ανταλλαγή απόψεων με τον αρμόδιο επίτροπο, τον κύριο Κάρλ Ντεχούχτ, τον οποίον καλώς ορίζω και πάλι, τακτικός ε, προσκεκλημένος εδώ στην επιτροπή μας. Και αυτή τη φορά ε, τον προσκαλέσαμε για να συζητήσουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, την πρωτοβουλία της Κομισιόν για ρύθμιση της λεγόμενου, του λεγόμενου μηχανισμού αμοιβαιότητας ε, δημοσίων προμηθειών. Δηλαδή, πρόσβαση των προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης, στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασίες που αποσκοπούν στη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων σχετικά με την πρόσβαση ε, των προϊόντων και υπηρεσιών της Ένωσης στην αγορά τρίτων χωρών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Δεν έρχεται συχνά ο κύριος Επίτροπος για συγκεκριμένο θέμα, αλλά αυτό το θέμα είναι βεβαίως πολύ σημαντικό. μα ενημέρωσε η Ιρλανδική Προεδρία πως είναι διχασμένο το Συμβούλιο, πως υπάρχουν πολλές επιφυλάξεις, πως πολλά κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα να μπουν σε συζήτηση για την πρόταση αυτή. Δεν υπάρχει λοιπόν αναθεωρημένη πρόταση του Συμβουλίου, οπότε η κατάσταση αυτή μου φαίνεται πως είναι μια κατάσταση η οποία απαιτεί να ακούσουμε την άποψη της Κομισιόν και να γίνουν κάποιες προσπάθειες παραπάνω για να ξεκαθαρίσει ε, την άποψή της. Η ε, Επιτροπή μας και ειδικά ο συγητής μας, ο κύριος Ντανιέλ Κάσφαρη, είναι αρμόδιος για αυτό το θέμα και βεβαίως αναμένουμε την άποψη του κύριου Επιτρόπου πάντα με ενδιαφέρον και αυτή τη φορά ε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω. Οπότε, καλώς ήρθατε και πάλι κύριε Επίτροπε. Στην Επιτροπή μας, την οποία μπορείτε να θεωρείτε σαν το σπίτι σας. Το σπίτι μου, ξέρετε, είναι μία φορά εδώ, μία φορά εκεί, λέει ο κύριος Επίτροπος μπορούσα να έχω και μία σκηνή να την πηγαίνω πέρα δόθε. Κύριε Πρόεδρε, και κύριοι βουλευτές, ξέρετε πως εγώ πιστεύω σε ανοιχτέ αγορές, Πιστεύω στην αμοιβαιότητα και ως Επίτροπος Εμπορίου θεωρώ πως βασικό καθήκον μου είναι να εργαστώ για το περαιτέρω άνοιγμα των αγορών για τις ευρωπαϊκές εταιρείες ο ευρωπαϊκός τομέας δημοσίων προμηθειών είναι από τους πιο ανοιχτού στον κόσμο και έτσι πρέπει να παραμείνει. Εταιρείε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι βεβαίως καλοδεχούμενες στο να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς μας ε, και βεβαίως αυτό δεν ισχύει παντού στον κόσμο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μόνο 5% των ε, διαγωνισμών που αφορούν ε, δίκτυα μετρό στους, δο, 12 μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους μας είναι ανοιχτές ε, σε ξένες εταιρείες. Και βέβαια έχουμε γύρω στα 350 δισεκατομμύρια δημόσιες προμήθειες που είναι ανοιχτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις χώρες με τις οποίες έχουμε ένα γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων. Αντιστρόφως όμως ε, οι... Στι χώρε αυτέ οι διαγωνισμοί στου οποίου έχουν πρόσβαση ευρωπαϊκέ εταιρείε έχουν ύψος μόνο 178 δισεκατομμυρίων. Στην Ιαπωνία δεν μόνο 7 δισεκατομμύρια. Βραζιλία και άλλες χώρες δεν έχουν ανοίξει καν τις ε, αγορέ του. Στι 28 Μαρτίου ε, προτείναμε κάποια μέσα την λεγόμενη διεθνή πρωτοβουλία δημοσίων προμηθειών για να υπάρξει ένας διεθνής συνταγωνισμός που θα ωφελήσει τις δουλειές και την ανάπτυξη. Η πρόταση αυτή προσπαθεί να βρει μια ισορροπία μεταξύ του να διατηρήσει ανοιχτέ τις ευρωπαϊκές αγορές δημοσίων προμηθειών και ε, να δίνει κάποιο μοχλό πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει τις ευρωπαϊκές εταιρείε. Και όπως αναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, οι απόψει των κρατών μελών είναι διχασμένες. Αρκετά κρατημέλη εξέφρασαν τις επιφυλάξεις τους ε, και ε, διαφωνούν πλήρες. πλήρως. Κάποια άλλα κρατημέλη ταυτόχρονα στήριξαν την πρωτοβουλία. Κατέθεσαν μάλιστα και συγκεκριμένες ε, πρωτοβουλίες ε, και προτάσεις τροποποίησης της πρότασης αυτής. Ελπίζω να γίνεται αντιληπτό πως ε, αποτελεί πρόβλημα το μία άνοιγμα των αγορών αυτών και θα πρέπει να διασφαλίσουμε και καλύτερη πρόσβαση των ευρωπαϊκών εταιριών σε τρίτες χώρες. Ειδικά καθώς οι δημόσιες προμήθειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μειώνονται λόγω λιτότητας και οικονομικής κρίσης. Όταν φτάσουμε στο ζήτημα του πώς πρέπει να αντιδράσει η Ένωση, εκεί πέρα αρχίζουν διαφωνίες. Κάποιοι λένε πως Θα πρέπει απλά να διατηρήσουμε το παρόν επίπεδο ανοίγματο και να προσπαθήσουμε για μεγαλύτερη πρόσβαση στις ξένες αγορές. Ε, οι διαδικασίες των ΠΟΕ έδειξαν πόσο δύσκολο είναι να καταλήξουμε σε δεσμεύσεις για πρόσβαση αγορές. Προφανώς σε διμερείς συμφωνίες υπάρχει κάποιο ε, περιθώριο ελιγμών γιατί είχαμε πρόσφατα αποτελέσματα σε τέτοιες συμφωνίες και σημειώνεται πρόοδος και στις διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Και βεβαίως θα ξεκινήσουν σύντομα διαπραγματεύσεις με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ. Αλλά βεβαίως διατομιακές τέτοιες συμφωνίες παραμένουν δύσκολες και δεν πρέπει οι εμπορικοί μας εταίροι να θεωρούν δεδομένο πως εμείς θα έχουμε ανοιχτές τις δικές μας αγορές και να αναζητούν και άλλες παραχωρήσεις ως αντάλλαγμα τα προτινόμενα μέσα παραμένουν μια σημαντική προσθήκη στα αυτά που έχουμε στην διάθεσή μας ήδη στις διμερείς διαπραγματεύσεις. Οι περιορισμοί στην πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά δημοσίων προμηθειών πρέπει να αντιμετωπιστούν στο ε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να έχουν διατάξεις ε, διακρίσεων ε, όσον αφορά τις δημόσιες προμήθειες, καθώς αυτές θα αντιβαίνουν το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η πρόκληση είναι ιδιαίτερα μεγάλη στις ε, αναδυόμενες οικονομίες όπου είναι πολύ πιο σημαντικές βραχυπρόθεσμα οι αγορές αυτές παρά το ότι βεβαίως είναι προς το συμφέρον τους να δουν τα πράγματα πιο ανοιχτά πράγματα. Χάρη ξεκάθαροι κανόνες δημοσίων προμηθειών σημαίνουν πως θα ε, υπάρξουν σημαντικές εξοικονομήσεις στις δημόσιες, στις δαπάνες. Και βεβαίως θα αντιμετωπιστεί έτσι και το ζήτημα της διαφθοράς και των δωροδοκιών. Πολλές χώρες αλλάζουν την άποψή τους. Η Ινδία και η Μαλαισία πρόσφατα έγιναν παρατηρητές στις σχετικές συμφωνίες του ΠΟΕ. Αλλά άλλες διστάζουν. Η Κίνα βεβαίω ε, χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να διαπραγματευτεί την ένταξή της στις ε, γενικές ε, στις γενικευμένες ε, προτιμήσεις. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε και την χρησιμότητα της πρότασης της Κομισιόν. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως πως ε, τα πράγματα είναι προκαθορισμένα. Πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία όπου θα εξετάσουμε τα διάφορα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και θα τα κρίνουμε. Και βεβαίως σκοπεύουμε να είναι όσο δυνατόν πιο ισορροπημένη και αποτελεσματική η διαδικασία και καλωσορίζω τις προτάσεις σας, όπως και αυτές του Συμβουλίου. Σύντομος και εύστοχος. Ευχαριστούμε κύριε Πίτροπε. Ας ανοίξουμε τη συζήτηση. Ο εισηγητής μας, κύριος Κασπάρη, ΕΛΚΑ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα. Είναι πράγματι εξαιρετικό να έρχεται ο Επίτροπος για να συζητήσει ένα συγκεκριμένο θέμα, αλλά για αυτό το συγκεκριμένο θέμα αξίζει. Σήμερα έχουμε την τρίτη τελεγγύη απόψεων για το θέμα, αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν τα εξή προβλήματα όταν μιλάμε με τους συναδέλφους εδώ στο Κοινοβούλιο, η εντύπωσή μου είναι πως υπάρχουν κάποιοι ήδη που απορρίπτουν τελείως την υπόθεση αυτή, αλλά το πρόβλημα είναι τα άρθρα 8 και 10. Και ε, το Κοινοβούλιο ασχεί κριτική στο άρθρο 6. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο έχουμε συζητήσει μόνο το άρθρο 6, οπότε από την άλλη στο Συμβούλιο μου λένε, αυτοί που είναι τελείως κατά αυτού του μέσου, που στο άρθρο 6 δεν τους δημιουργεί πρόβλημα. Τα βασικά τους προβλήματα εκεί πέρα είναι τα άρθρα 8 και 10. Και θα είμαι σαφής. Ερχόμαστε τώρα στο θέμα στο οποίο πρέπει να υποβάλω το σχέδιο έκθεσής μου, αλλά δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω από εδώ και μπρος για να εγκριθεί η έκθεσή μου. Γιατί Εμείς είμαστε υπέρ ενός μέσου που θα επεκτείνει και θα ενισχύει τα άρθρα 8 και 10, αυτά δηλαδή τα οποία είναι ακριβώς απαράδεκτα για το Συμβούλιο. Τι θα κάνουμε λοιπόν. Και το ερώτημά μου προς εσάς, προς την Κομισιόν, είναι αν έχετε καμιά ιδέα για να επιλύσουμε αυτή τη διαφωνία. Γιατί δεν χρειάζονται μεγάλα λόγια. Το θέμα είναι τι προοπτικές έχουμε για να ε, ξεπεράσουμε αυτή τη διαφωνία και την ε, ε, μειοψηφία που μπλοκάρει τα πράγματα στο Συμβούλιο. Γιατί αυτά τα οποία θέλουμε εμείς στο ε, Κοινοβούλιο είναι απαράδεκτα για το Συμβούλιο. Οπότε το ερώτημά μου είναι, έχετε κάποια στρατηγική, έχετε κάποια συμβουλή να μας δώσετε, τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο αυτό. Ευχαριστώ. Εγώ αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κασπαρή είναι ποια πιστεύετε εσείς ότι είναι η λύση, γιατί είστε εισηγητής μόνο. Ε. Ναι, σας ρωτάει. Αλλά και εγώ μπορώ να κάνω μια ερώτηση στον κύριο εισηγητή. Λέει, μιλάει για συμβατότητες και κάποιους που είναι υπέρ της λύσης Α, άλλοι της λύσης Β και πρέπει να λύσουμε αυτό το δεσμό, αυτό το γόρδιο δεσμό. Ίσως να έχετε κι εσείς κάτι να προτείνετε ή αλλιώ μπορείτε να μας πείτε δεν έχω κάποια άποψη, δεν θέλω να έχω άποψη, αλλά αν έχετε κάποια άποψη θα ήθελα να την ακούσω. Αν έχετε κάποια άποψη για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Καλά, εύκολο είναι να ανταλλάσσουμε ερωτήσεις, αλλά αυτό δεν βοηθάει ιδιαίτερα. Και αν θυμάμαι καλά, αυτή δεν ήταν πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι μια ιδέα παρουσίασε η Κομισιόν. Αποτελεί λοιπόν στο ευθύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας πει πώς θα υλοποιήσουμε τα έργα και αποτελεί καθήκον του κυρίου Σιγητή να βεβαιωθεί ότι θα λάβουμε πλειοψηφία στο κοινοβούλιο για κάτι και αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η πλειοψηφία που βλέπω σε... για αυτό το έργο στο κοινοβούλιο οδηγεί προ ε, έναν δρόμο που θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα με το Συμβούλιο διότι στο Κοινοβούλιο υποστηρίζουμε τα άρθρα 8 και 10 σε μεγάλο βαθμό και βλέπουμε προβλήματα με το άρθρο 6 και στο Συμβούλιο σημαίνει το ακριβώς αντίστροφο. Και η ερώτησή μου είναι ότι μήπως την ημέρα που θα παρέχουμε κάτι, θα παρέχουμε κάτι που θα βαίνει προς ποια κατεύθυνση. Και η ερώτησή μου είναι εσείς ως ε, πηγή αυτής της πρότασης. Είμαστε εδώ για να σας υποστηρίξουμε, να σας ελέγχουμε, αλλά όχι για να επιλύσουμε τα δικά σας προβλήματα. Πιστεύω αποτελεί πρόβλημα της Κομισιόν η Κομισιόν είναι εκείνη που πρέπει να μας βοηθήσει να επιτύχουμε πλειοψηφία για αυτή την πρόταση. Ναι. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις, αλλά θα μείνω όσο θέλετε, λέει ο Επίτροπος. Η ιδέα σας ότι δεν είστε εδώ για να λύσετε τα προβλήματα της Κομισιόν με εκπλήσει. Νομίζω ότι είχαμε την νομοθετική πρωτοβουλία εμείς και ότι εσείς στη συνέχεια έχετε ένα διτό σύστημα μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για να καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Όταν μου λέτε λοιπόν ότι δεν είμαστε εδώ για να λύσουμε τα προβλήματά σας, εμείς κάνουμε προτάσεις και είμαστε διαδεθμένοι να τις συζητήσουμε μαζί σας. Πολύ περίεργη αυτή η προσέγγιση του νομοθέτη που είστε. Θα προσπαθήσω να σας ε, παρουσιάσω μια λύση στο τέλος, αλλά ε, το να μου λέτε ότι δεν είμαι εδώ για να λύσω τα δικά σας προβλήματα, εγώ δεν έχω προβλήματα, ήρθα να σας κάνω μια πρόταση. Ως πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, μου επιτρέπετε να πω και εγώ τη δική μου άποψη. Αρμόζει απόλυτα για αυτό το κοινοβούλιο όταν έχει να κάνει με μια πρωτοβουλία της Κομισιόν η οποία φυσικά θέλει η πρωτοβουλία της να υιοθετηθεί σε αυτό το κοινοβούλιο και εμείς ε, δυσκολευόμαστε κατά την εξέτασή σας, είναι λογικό να ζητήσουμε βοήθεια από την Κομισιόν για να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Πιστεύω λοιπόν ότι η ερώτηση του κυρίου ε, Κασπάρη είναι απολύτως σωστή. Ο επόμενος ομιλητής θα ήταν ο κ. αλλά δεν είναι εδώ γιατί εξελέγει στο Ιταλικό Κοινοβούλιο και θα τον αντικαταστήσει ο Μπετλάνγκη από το S&D. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ διαφωνώ κάπως με τον κύριο Κασπάρη. Η αναγκαιότητα ενός τέτοιου μέσου έχει διατυπωθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, οπότε πρέπει να προωθήσουμε την ομοθετική διαδικασία. Ο λόγος για τον οποίο θέλουμε μια κοινή προσέγγιση υπάρχει. Και τα έχει ξεκαθαρίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οπότε πρέπει να δούμε τώρα τι θα κάνουμε με την κατάσταση που έχουμε μπροστά μας. Να δούμε ποιες είναι οι αντιστάσεις που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη. Εάν πέρα από τα βιολογικά ζητήματα που κάποιοι θεωρούν πως ε, υπάρχει πρόβλημα με την ελεύθερη αγορά, εντάξει δεν μπορούμε να τα λύσουμε, αλλά υπάρχουν κάποια πράγματα δικαιολογημένα τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Το ένα είναι ο διοικητικός ε, φόρτος, ειδικά στο τοπικό επίπεδο. Αυτό μπορούμε να το ελαχιστοποιήσουμε ειδικά σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα όπως η Γερμανία, μπορεί ε, για τις τοπικές αρχές να σημαίνει κάτι τέτοιο περισσότερο.